So, I'm so sorry. Good afternoon, everybody. Καλό από μεσήμερο. Ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα το απόγευμα ανάμεσά μας. Συγγνώμη για την λαφρά καθυστέρηση απελπισμένα αναζητούσα την ηλεκτρονική μου κάρτα πρωτού σας ε, ζητήσω να έχετε τις δικές σας αλλά δυστυχώς ε, δεν ε, βρέθηκε, δεν ξέρω τι έκανα με την τελευταία μου ηλεκτρονική κάρτα ζήτησα σε κάποιον να έρθει να μου την φέρει είναι απαραίτητο, θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η έγκριση της ημερησίας διατάξεως αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνεται ως 8 τη μέσα διάταξη. Και τώρα περνάμε σε ανακοινώσει του Προέδρου. Θέλω να σας ζητήσω να, να στηρίξετε τις συστάσεις των ε, συντονιστών για τα παρακάτω θέματα και εισηγητές πρώτον γνωμοδότηση για τον προβλησμό 2017 εισηγητής ο κ. Γιακολίνο γνωμοδότηση για την πρόγραμμα για Ευρώπη περί των πολιτών, εισηγητής ε, κ. Σάμπα Σόγκουρ. Τρίτον, έκθεση πρωτοβουλία ε, όπως ζήτησε η Ολομέλεια ε, το ψήφισμα τον Φεβράριο του 2012, ο κ. Ρούι Ταβάρες, εισηγητής, γνωμοδότηση για το ζήτημα των προσώπων που κατέχουν πληροφορίε και για πράξη χειραγώγη αγορά ε, ε, κυρία ε, δεν υπάρχουν λοιπόν ενστάσει, εγκρίνονται οι συστάσει αυτέ. Αναγγέλλω επίση πω την ε, πρόσφατο Συμβούλιο ΔΕΗ, μάλλον στο επόμενο Συμβούλιο, συγγνώμη, στο Συμβούλιο του Μαρτίου, Αυγούστος ενεκρίθη ε, έκθεση για την ε, αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη που υφίστανται πιέσεις σε ό,τι φορά τη χορήγηση ασύλου για τα μεικτά μεταναστευτικά ρεύματα. Το πλαίσιο θεωρείται ως ευέλικτο και ανοιχτό ε, ανοιχτή εργαλειοθήκη που συνδυάζει τα εφιστάμενα και τα πιθανά νέα μέτρα που θα αφορούν ε, την ε, αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τους ε, ετούντε άσυλο και από τα μεικτά μεταναστευτικά ρεύματα μετά, ως απάντηση μετά από αίτημα της Κομισιόν για την ενδονοσιακή αλληλεγγύη. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αύριο στην συνεδρίασή μας. Αυτές είναι οι αναγγελίες και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την νημιστή η οποία περιλαμβάνει κάποια σημαντικά σημεία αλλά προηγούμενα αλλά υπάρχει ανακοίνωση σχετικά με την προστασία δεδομένων. Γνωρίζετε ότι η έκθεση περί προσωπικών δεδομένων συζητήθηκε τουλάχιστον σε τρεις συνεδριάσεις των συντονιστών. Στην τρίτη συνάντηση που διεξήχθη την 7η Μαρτίου, η πλειοψηφία των συντονιστών επιβεβαίωσαν τις ε, εκθέσεις, δύο εκθέσεις ε, περί του θέματος ε, που εμπλέκουν και το λεγόμενο point system. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν ο... το θέμα ανατέθηκε στους πρασίνους και η οδηγία στην ομάδα των σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών. Ο... Το άρθρο 192 του κανονισμού αναφέρει και παραθέτω ότι συντονιστές θα πρέπει να προσπαθούν να βρουν συνένεση. Όταν η συνένεση δεν είναι δυνατόν επιτευχθεί, τότε μπορούν να ενεργήσουν με την πλειοψηφία που αποτελεί την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία της Επιτροπής και λαμβάνει υπόψη την δύναμη των, πολιτικών ομάδων. Αυτή η συνεδρία των συντονιστών που έλαβε χώρα την 7η Μαρτίου ε, σε αυτή την ομάδα αφισβήτησε το ΕΛΚ ως εκ τούτου η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε τα συμπεφωνημένα από την συνεδρίαση των συντονιστών θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολο της Επιτροπής ε, προς ψήφιση. Η διάσκεψη των Προέδρων που εκλήθη να εξετάσει το θέμα στη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου συζήτησε την υπόθεση και παραθέτω εκ νέου ότι ζήτησε από τους συντονιστές να εξεύρουν μια συνενετική λύση στο πλαίσιο της, ομάδας, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως το ΕΛΚ ζήτησε μια μετάθεση της ψηφοφορία και αυτό θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για τις πιθανότητες που έχουμε να βρούμε μια συνενετική λύση με την ανάθεση των εκθέσεων και έχουμε και μια σειρά από πολιτικές ομάδες οι οποίες όμως επέμειναν στο να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του θέματος όπως ε, είχε συμφωνηθεί στη συνεδρίαση των συντονιστών ε, την 7η Μαρτίου. Ούτε συγχώνων των πραγμάτων λοιπόν προτείνω να έχουμε δύο ε, ψηφοφορίες. Η πρώτη θα την προηγούμενη προηγούμενη απόφαση, δηλαδή είμαστε, είσαστε έτοιμοι να ψηφίσετε σήμερα ή θα προτιμούσατε να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με την πρόταση του ΕΛΚ. Στην περίπτωση αυτή θα μεταθέσουμε την ψηφοφορία και θα διεξαχθεί στην προσεχή συνεδρία της Βουλής Λίμπε 26 Μαρτίου στις 15.00. 26 Μαρτίου, 3 το απόγευμα λοιπόν, θα ψηφίσουμε επί του θέματος. Αλλά στην περίπτωση που ψηφίσουμε σήμερα δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε ειδικά με την ε, ανάθεση των ανωτέρων εκθέσεων η ερώτηση θα έχει οξύ. Εγκρίνεται ή όχι την απόφαση των συντονιστών της 7ης Μαρτίου. Λοιπόν, εάν μου κατέστη τη σαφή, εάν τα είπα σωστά με άλλα λόγια, θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, η οχι την αποφαση των συντονιστων της 7 ης μαρτιου λοιπον εαν κατεστη την σαφη εαν τα ειπα σωστα με αλλα λογια θα ψηφισουμε λοιπον η αποφαση 1 συμφωνούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Ψηφίζουμε σήμερα το θέμα της ανάθεσης των εκθέσεων. Αυτό θα ψηφίσουμε πρωτίστως. Άρχεται η ψηφοφορία και προτείνω για να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Λοιπόν, συμφωνείτε να ψηφίσουμε τώρα ή θέλετε μετάθεση. Αν συμφωνείτε για σήμερα θα ψηφίσετε ναι. Αν ε, δεν συμφωνείτε θα ψηφίσετε όχι. What is it? I have report. Μου λένε εδώ ότι περισσεύουν τρία μέλη του ΕΛΚ. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό. Και επίσης περισσεύει και ένας σοσιαλιστής δημοκράτης. Όχι, έχει εξαφανιστεί ο σοσιαλιστής. Αλλά περισσεύουν τρεις ψήφοι του ΕΛΚ. Τρεις ψηφίζουν χωρίς να δικαιούνται. Εντάξει, εντάξει, τα βρήκαμε. Ψηφίστε τώρα. Όχι, ένας του ΕΛΚ πρέπει να αποσυρθεί. Εντάξει, ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πάλι δεν έχει αποσυρθεί μία ψήφος του ΕΛΚ που περισσεύει. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 25 κατά, άρα θα ψηφίσουμε τελικά. Θα ψηφίσουμε για την κατάνομή των εκθέσεων. 31 ψήφισαν υπέρ, 25 κατά, κανένας δεν απήχε. Οπότε θα ψηφίσουμε. Τώρα, θα εγκρίνουμε ή όχι τις συστάσεις των ε, συντονιστών για τις δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας, την προστασία δεδομένων, ε, τον κανονισμό στους πράσινους και την οδηγία στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ψηφίζουμε για το κατά πόσο θα εγκρίνουμε την απόφαση των συντονισμών. Διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε, για όσου απουσίαζαν από την ε, συνεδρία των συντονιστών, θα ήθελα να πω ότι η θέση του ΕΛΚ σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί τη χρήση του συστήματος με, τα, με τους πόντους. Η έκθεση αυτή, για την οποία ψηφίζουμε, είναι μια έκθεση για την οποία είχαμε εκδηλώσει ενδιαφέρον τον Ιανουάριο του 2011, όχι φέτος, πέρυσι, τον Ιανουάριο του 2011, Δυστυχώ δεν χρησιμοποιούσαμε τότε το σύστημα των πόντων, αλλά έγινε κατάχρηση του συστήματος αυτού για μια ολόκληρη χρονιά. Γι' αυτό και ζητήσαμε σήμερα διαδικαστική ψηφοφορία. Δεν πρόκειται για επίθεση κατά του συστήματος των πόντων, αλλά θέλουμε μια πιο συνενετική κατανομή των διαφόρων εκθέσεων. Καλώς ακούσαμε μια εκτενή ε, εξήγηση της θέσης του ΕΛ και του γιατί ζητήθηκε ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα την ανάθεση των εκθέσεων. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Και πάλι περισσεύει μια ψήφος του ΕΛΚ. 32 δύο υπέρ, 26 κατά. Χωρίς αποχές, άρα εγκρίνεται η πρόταση για την ανάθεση των εκθέσεων με βάση το σύστημα των πόντων. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην κανονική μας ημερήσια διάταξη και σας ευχαριστώ όσους ε, ήρθαν εγκαίρως για την ψηφοφορία. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε, κάνοντας λίγη ησυχία, Again, dear colleagues, please those leaving the room. Συνάδελφοι, παρακαλώ, όσοι αποχωρούν από την αίθουσα, να μην κάνουν φασαρία για να μην εμποδίσουν την συνέχεια των εργασιών. Είπα ησυχία. Help us. After Mrs. Wikström wanted to take the floor after the after the vote. Yes, yes, yes. We are ready to get started with the agenda. We have a full agenda. Έχουμε μία πληρέστατη ημέρη σε διάταξη. Οπότε χρόνου φίδου. Η κυρία Βίξτρομ ζήτησε το λόγο για να εξηγήσει την ψήφα της όμως. Όχι καθόλου, καμία σχέση. Δεν θέλω να εξηγήσω την ψήφα μου. Άλλο είναι το ζήτημα που θέλω να θίξω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο πέντε μεταναστών το προηγούμενο Σαββατοκυριακό που έχασαν τη ζωή τους ε, στην ε, Μεσόγειο προσπαθώντας να φύγουν από τη Λιβύη και να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Σικελίας. Μερικοί έφτασαν, κατάφεραν και αυτά στη Λαπεντούζα, άλλοι θα επαναπατριστούν ε, πάραφτα από τη Μάλτα και την Ιταλία εξαιτίας του κλεισίματος του λιμανιού της Λαμπεντούσα Φαίνεται λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι ξαναζούμε σκηνές του παρελθόντος με ανθρώπους να πνίγονται στη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε ότι πέρσι η αποστολή της Επιτροπής μας πήγε στην Σικελία. Ήμουν επικεφαλής αντιπροσωπείας και επισκεφτήκαμε τότε μερικούς καταφλισμούς προσφύγων ε, μεταναστών, δηλαδή, συγγνώμη, στο νησί. Και συζητήσαμε πολλά και διάφορα θέματα με τις τελικές αρχές, που περιέχοντας σε μια επιστολή που είχα στείλει στις τελικές αρχές, ζητώντα πιο διεξοδικές πληροφορίες για την διακήρυξη της Λαπεντούσα ως ε, ε, μη ασφαλές λιμάνι για τους μετανάστες, αλλά ασφαλές για τους αλληλείς και τους τουρίστες. Παρά τις υποσχέσεις των Ιταλικών αρχών, ότι έστειλαν απάντηση. Εγώ για πολύ καιρό δεν έλαβα τίποτα. Πέρασαν δύο μήνες και εν αναμονή της απάντησης των Ιταλικών αρχών. Ε, θα ήθελα να απευθύνω λοιπόν έκκληση προς τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπή αυτή να καταθέσουμε μία προφορική ερώτηση ζητώντας από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν δράση. Αυτό θα κάνω τουλάχιστον εγώ εκ μέρους της δικής μου πολιτικής ομάδας. Στόχος της προφορικής αυτής ερώτησης είναι να εξασφαλίσουμε σωστή ε, μεταχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προστασία των ε, ε, των τον από επαναπατρισμό ή πνιγμό στη θάλασσα. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα υποστηρίξουν την προφορική μου ερώτηση και σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ναι, συμφωνούμε κύριε Βίξτρομ μαζί σας και σε ευχαριστούμε για τη δήλωση. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό όντως. Και βλέπω ότι ζήτησε το λόγο ο κύριος Μπρόγκς για το ίδιο θέμα. Παρακαλώ να είστε λακωνικός. Ναι, συμμερίζομαι και εγώ την θλίψη της κυρίας της ε, Wickstrom για την τραγωδία αυτή, το πνιγμό. Θα... Την είχαμε όμως αποφύγει ίσως, αν μπορούσαμε να εξηγήσουμε σε όλους τους κατοίκους της Λιβύης ότι η δημοκρατία έχει φτάσει πια στην πατρίδα τους και ήρθε η ώρα να παραμείνουν στη χώρα τους και να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της δημοκρατίας και όχι να προσπαθούν να φύγουν μακριά από τη δημοκρατία. κυρία Wickstrom σε ολόκληρη τη Μεσόγειο μόνο δύο λιμάνια θεωρούνται ε, μη ασφαλή. Είναι της Λιβύης και της Λαμπεντούζα. Αυτή ήταν η δήλωση της α, την οποία ηγήθηκα, της οποίας ηγήθηκα πέρυσι. Ας μην ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Θα στείλω την προφορική ερώτηση στα μέλη της αντιπροσωπείας το συντομότερο δυνατόν. Καλά, ας μην αρχίσουμε τώρα συζήτηση. Το θέμα αυτό δεν είχε προβλεφθεί στην ημερήσια διάταξη. Αν, ας μην την φορτώνουμε με επιπλέον σημεία γιατί ήδη είναι κατάμεστη. Έχουμε πέντε θέματα και μόνο τρεις ώρες και δέκα λεπτά για να τα διεκπαιρεώσουμε. Προσοχή λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια πολύ ορθολογική κατανομή του χρόνου. Το σημείο 4. Γενικέ διατάξει. Ταμείο για το άσυλο και τη μετανάστευση και μέσω χρηματοδοτική στήριξη. Πρόκειται για την έκθεση Λορέντζο Φοντάνα. Προβλέπεται παρουσίαση από την Επιτροπή και πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Με την περίοδο 2014 ε, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και τον κανονισμό που αφορά τη χρηματοδότηση, τους τρόπους ε, της χρηματοδότησης την, έγκριση, την ε, κατάρτιση και έγκριση των εθνικών προγραμμάτων και το καθεξής. Περιμένουμε λοιπόν ε, την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την παρουσίαση. Μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή μας τον κύριο Φοντάν από την Ευρώπη της Δημοκρατίας και Ελευθερίας και θα γίνει και συζήτηση. Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα αφιερώσουμε μισή ώρα σε αυτό το πρώτο σημείο της απογευματινής ημέρη διάταξης. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκπρόσωπο μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μπελίντα Πάικ και την παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα θέματα 4 έως 7 συνδέονται μεταξύ τους. Ε, αποτελούν το πακέτο εσωτερικών ε, θεμάτων ε, και το πολιτές ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Γενικός μου Διευθυντής ήρθε στην Επιτροπή σας στις 29 ε, Σεπτεμβρίου να σας παρουσιάσει την πρόταση της Κομισιόν. Τότε τα κείμενα δεν ήταν διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Εκτιμούμε ότι αυτή είναι η πρώτη δυνατότητα που έχουμε να συζητήσουμε τις προτάσεις μαζί σας με βάση το νομοθετικό κείμενο. Ήδη έχουμε στείλει στην γραμματεία για να διανύμει στους ευρωβουλευτές ε, κάποιες πληροφορίες. Καταρχήν ε, μια σειρά διαφανειών ε, που ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμες ως πληροφορίες. Επίσης έχουμε στείλει κάποια ενημερωτικά φυλάδια τα οποία είχαμε ετοιμάσει για να βοηθηθεί η συζήτηση που είχε ήδη ξεκινήσει στο Συμβούλιο. Ήδη έχουμε παρουσιάσει στο Συμβούλιο και τώρα πια και στη ΛΥΜΠΕ έξι τέτοια φυλάδια τα οποία εξηγούν κάποια από τα στοιχεία ε, των προτάσεων αυτών. Και Ευχαρίστω θα σα στείλουμε και οποιοδήποτε άλλο φυλάδιο που θα στείλουμε και στο Συμβούλιο. Να σα ε, πω για τι ε, συζητήσει ε, στο Συμβούλιο ότι έχει δημιουργηθεί μια ομάδα ad hoc τώρα υπό την Δανική Προεδρία για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Είναι η ίδια ομάδα που ασχολείται και με τι προτάσει δικαιοσύνη, αλλά ιδιαίτερα για το πακέτο εσωτερικών και άλλωστε έχουμε εκπρόσωπο του Συμβουλίου εδώ. Προχωράμε σε κάθε ένα από τα θέματα αυτά. είναι λοιπόν και το Συμβούλιο παρόν και θα μπορείς να ακούσει αυτά που έχουν να πούν οι ευρωβουλευτές Να σα θυμίσω ότι οι δαπάνε ε, για τα θέματα εσωτερικού ε, στα πλαίσια του πολιετού ε, δημοσιονομικού πλαισίου αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 1%. Το ίδιο προβλέπεται για το μέλλον, αλλά γενικά αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση τάξεως του 40% και αυτό αντικατοπτρίζει την σημασία που δίδεται στις ε, πολιτικές εσωτερικών. Το ε, χρηματοδοτικό πακέτο για τα θέματα εσωτερικών ε, προβλέπει δαπάνες και για τους σχετικούς οργανισμούς και για τα συστήματα πληροφορικής που ήδη έχουν ε, αναπτυχθεί ε, και που βρίσκονται στο τελικό τους ε, στάδιο. Το σύστημα Schengen 2, το σύστημα πληροφόρηση Schengen 2, το Eurodac και άλλα. Και φυσικά μόλις έχει δημιουργηθεί ο Οργανισμός Πληροφορικής για τη διαχείριση των συστημάτων αυτών. Στη σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθούμε κυρίως στα δύο νέα ταμεία αυτό για το άσυλο και τη μετανάστευση και αυτό για την εσωτερική ασφάλεια. Θα ήθελα να συνοψίσω την γενική ε, προσέγγιση προτού να μιλήσω σύντομα για το πρώτο μέσο από το οποίο συζητάμε τώρα. Γενικά προβλέπουμε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για ε, τα δύο αυτά σημαντικά ταμεία. Οι εμπειρίε από το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι θετικές, ε, αλλά υπάρχουν ε, περιορισμοί όσον αφορά τους τύπους των μέσων που έχουμε και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, σε επίπεδο εσωτερικών. Κάποια από αυτά μόλι μα τα θύμισε η κυρία Βίξτρομ. Ε, έχουμε δύο ξεχωριστά ταμεία και δύο προγράμματα. Ε, σκοπός ε, στο μέλλον είναι να έχουμε δύο ταμεία, το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας με έναν μηχανισμό όμως. Και αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε ε, σε αυτό το θέμα τη ημερήσια διάταξη είναι ακριβώ αυτό ο μηχανισμό. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, διαβάσουμε τα διάφορα κείμενα χωρί να έχουμε κατά νου ότι ο μηχανισμό ε, περιγράφεται στον κανονισμό στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για τα ταμεία αυτά, τα 2 τρίτα θα ταπανώνται με κοινή διαχείριση σε εθνικά προγράμματα κατόπιν συμφωνίε με τα κράτη-μέλη σε πολυετή βάση. Μπορεί να Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή τα εθνικά προγράμματα συμφωνούνται σε ετήσια βάση το οποίο επιβάλλει κάποιους περιορισμούς. Ε, τα περισσότερα από τα χρήματα στα προγράμματα αυτά θα κατανεμηθούν ε, στην αρχή του, του διαστήματος ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το μεγαλύτερο μέρος με βάση ένα συγκεκριμένο, ένα βασικό ποσό, θα σας το εξηγήσουμε αυτό όταν φτάσουμε στα επιμέρους μέσα, και κάποια χρήματα θα δοθούν Ε, για να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε, κάποια, σε κάποιους τύπους δράσεων. Ε, όταν μιλάμε για το Ταμείο για το και τη Μετανάστευση και για το Ταμείο ε, Εσωτερικής Ασφάλειας, ε, θα σας ε, εξηγήσουμε ποια είναι αυτά τα μέσα. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα 2017 να γίνει ενδιάμεση αναθεώρηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ε, περαιτέρω ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων για να ληφθούν υπόψη θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση στην εσωτερική ασφάλεια. Τα δύο τρίτα λοιπόν ε, του ποσού θα ε, δίδεται με κοινή διαχείριση, ενώ το ένα τρίτο θα δίδεται με άμεση διαχείριση ε, για δράσεις σε τρίτες χώρες μεταξύ άλλων. Το θέμα της άμεσης διαχείρισης ε, θα σας το εξηγήσω όταν φτάσουμε στο Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια για τα σύνορα. Θα σα εξηγήσω το θέμα ε, των ε, ευφυών σύνορων και αυτό θα αποτελεί αντικείμενο άμεσης διαχείρισης. Γιατί έχουμε διάφορα μέσα. Νομίζω ότι ο Γενικός μου Διευθυντής στα τέλη Νοεμβρίου σα το εξήγησε αυτό. Ε, υπάρχουν λόγοι που έχουν να κάνουν με τη συνθήκη. Ε, και γι' αυτό ε, ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε τρία κάθετα μέσα. Έχουμε το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και κατόπιν ε, έχουμε το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια για την Αστυνομία και το Ταμείο για την Εξωτερική Ασφάλεια, Εξωτερικά Σύνορα και Θεωρήσει. Δύο σκέλη δηλαδή για το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια. Έχουν όμω ένα κοινό στοιχείο που είναι το κοινό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο αυτού του θέματο στη μέση διάταξη. Επιτρέψτε μου σύντομα να συνοψίσω τα πλεονεκτήματα αυτού του οριζοντίου ε, μέσου. Καταρχήν αποφεύγουμε επικάλυψη μεταξύ των ταμείων. Δεύτερον, έχουμε έτσι απλοποίηση και συνέπεια, διότι οι ίδιοι κανόνες θα ισχύουν για όλους τους δικαιούχους. Ε, έτσι λοιπόν βελτιώνεται η κατανόηση από πλευρά των κρατών μελών και άλλων δικαιούχων ε, σχετικά με το πώς λειτουργούν τα ταμεία αυτά και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα βελτιώσει την πρόσβαση στα ταμεία. Και τρίτον, έχουμε μια ε, πιο ευθεία προσέγγιση ε, σε θέματα ε, εσωτερικών. Για παράδειγμα, θα έχουμε έναν ενιαίο διάλογο με τα κράτη-μέλη για τη χρηματοδότηση των κρατών μελών για το διάστημα της επταετίας στα θέματα εσωτερικών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτού του κανονισμού πλαισίου που συζητάμε τώρα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να επιστήσω την προσοχή σας στην κοινή διαχείριση και την προσέγγιση του προγραμματισμού. Εδώ υπάρχουν δύο ε, ιδιότητες που νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή σας. Καταρχήν έχουμε την εταιρική σχέση, την αρχή της εταιρική σχέσης, η οποία υπήρχε στις υπάρχουσες διατάξεις, δεν ε, έχει αναπτυχθεί όμως στον ίδιο βαθμό με άλλους τομείς ε, κοινοτικής ε, χρηματοδότησης. Θέλουμε λοιπόν σε συνεργασία με τους σχετικούς παράγοντες ε, να ε, εξετάσουμε την πτυχή αυτή και επίσης το άλλο σημαντικό είναι ο πολιτικός διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος που θα πραγματοποιηθεί μάλλον το 2013 και θα είναι μια ευκαιρία για το κράτος μέλος και την Κομισιό να συμφωνήσουν ποια ε, θα είναι η βάση στο κράτος μέλος αυτό και ποιος θα είναι ο στόχος της χρηματοδότησης. Μετά από τον πολιτικό αυτό διάλογο που θα επιβεβαιώνεται με ε, πρακτικά ή με ανταλλαγή επιστολών. Ε, το ε, λόγο κράτος μέλος κατόπιν θα στέλνει το πολιετές του πρόγραμμα. Θα υπάρχει ένα πρόγραμμα για το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και ένα για το Ταμείο για την Εστερική Ασφάλεια. Τα άλλα θέματα στα οποία θα ήθελα να την προσοχή σας μέσα στον κανονισμό αυτό είναι ότι όσον αφορά τον ε, χρηματοοικονομικό ε, έλεγχο, κάποιες ε, διατάξεις πήραν, τις εμπνευστήκαμε από άλλες διατάξεις σε άλλους τομείς. Έχουμε όμως εφαρμόσει αναλογική προσέγγιση. Τα οι ευρωβουλευτές έχουν λάβει λεπτομέρειες, ε, οι ε, σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο. Ε, δεν χρειάζεται να εμβαθύνω σε αυτά. Ευχαριστώ όμω θα απαντήσω στις σχετικές ερωτήσεις. να αναφερθώ στον συγκεντρωμένο τρόπο διαχείρισης που θα είναι κάτι που θα δείτε και στις παρουσιάσεις του ε, Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και του Ταμείου για την Εσωτερική Ασφάλεια έχει να κάνει με τη δυνατότητα να δαπανούμε χρήματα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι πολιτικέ εσωτερικών που έχουν και εξωτερική διάσταση. Ε, για του τομεί αυτού θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δαπανώνται χρήματα σε τρίτε χώρε. Έχουμε εργαστεί πολύ προσεκτικά όμω για να φροντίσουμε να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στη χρηματοδότηση με εξωτερικά μέσα. Δεν Πρόκειται για δράσεις οι οποίες στόχο έχουν ε, να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται ε, για εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Το βασικό μου μήνυμα είναι πάντως ότι αυτό είναι ο κανονισμός πλαίσιο ο οποίος διασφαλίζει το περιεχόμενο των σχετικών κανονισμών για το μείο την εσωτερική ασφάλεια και το άσυλο και τη μετανάστευση. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Λορέντσο Φοντάνα, παρακαλώ εν συντομία. Δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος από το Συμβούλιο να λάβει το λόγο. Πολύ ευχαριστώ. Είναι πρόσδεκτη η Δανική Προεδρία να λάβει το λόγο. Η κυρία Σίτσερ Μίλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για τη συνάντηση αυτή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να συναντηθώ και με τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές. Θα είμαι λακωνική, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όπως ανέφερε και η κυρία Μπελίντα Πάικ, ότι συστήθηκε μια ad hoc ομάδα του Συμβουλίου για τη διαπραγμάτευση των χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά για την περίοδο 2014-2020. Εγώ είμαι πρόεδρος αυτής της ομάδας εργασίας για τις εσωτερικές υποθέσεις που έχει αναλάβει την εντολή να διεξαγάγει διαπραγματεύσει για αυτά τα τέσσερα χρηματοδοτικά μέσα που εξετάζουμε σήμερα. Η Κορεπέρ σύστησε στις 10 Ιανουαρίου του 2010 αυτή την ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας ενημερώνει απευθεία την Κορεπέρ, αλλά θα, θα ενημερώνει και τα, α, τις ομάδες εργασίας Κάτς, Κίφα, κουσί και Τζάετς. Παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις για το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020 και γι' αυτό συζητούμε μόνο τα αριθμητικά στοιχεία. Η Προεδρία θα υποβα... Ε, ασχολείται με τις προτάσεις ως, ως, πακέτο. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια ολιστική συνολική προσέγγιση είναι χρήσιμη και συνάδει με την πρόταση ανασυγκρότησης των ταμείων. Θέλουμε να σημειωθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη πρόοδος για αυτό το, το συνδυασμένο ταμείο και έχουμε προβλέψει περίπου 16 συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση γιατί σήμερα δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα εργασίες και έτσι δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Στο μέλλον όμως θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για πιο διεξοδική ενημέρωση. Πάντως ε, θα παρακολουθήσουμε ιδιαίτερη προσοχή τη συζήτηση και τα σχόλιά σας. Ωραία. Ο εισηγητής μας τώρα, ο κύριος Λορέντσο Φοντάνα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Κομισιόν για την έκθεσή της θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβω καλύτερα ποια είναι τα κριτήρια που θέλουν να υλοποιηθούν. μίλους για τρίτα κράτη. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς πιστεύει ότι μπορούν να ελεγχθούν αυτά τα κονδύλια που θα χορηγούν σε τρίτες χώρε γιατί αυτό της εποπτείας, ε, της παρακολούθησης ε, με ανησυχεί όχι μόνο για τις τρίτες χώρες αλλά και για τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, γνωρίζουμε πως δυστυχώς ε, συχνά τα ταμεία χρησιμοποιούνται με τρόπο εσφαλμένο ή δεν χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε αν ε, μήπως και μέσω πρόθεσμα δεν είναι ε, μια προθεσμία πολύ μακρινή. Ακόμα και αν είναι πολύ τα προγράμματα, ειδικά ε, σε ό,τι φορά τις χώρες που είχαν προβλήματα στο παρελθόν. Ένας κάποιος έλεγχος, μια κάποια παρακολούθηση δεν θα ήταν κακό. Κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω αφορά την βοήθεια σε καταστάσεις επίγουσες. Ε, γνωρίζουμε δυστυχώ πω ορισμένε φορές υπάρχουν κατεπήγοντα συμβάντα όπως συνέβη και πάνω από ένα έτος ε, με την Αραβική Άνοιξη που οδήγησε σε μια αύξηση της μετανάστευσης από τις χώρες αυτές. Πολλά κρατημέρια αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίε. Διερωτώ με λοιπόν, ε, επειδή δυστυχώ τότε είχα ε, ακούσει ότι οι ε, ορισμένες χώρες είχαν εγκαταλειφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέλω να γνωρίζω εάν προβλέπετε κάτι για να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν για κάποια κράτη. Ε, αυτά ως ερωτήσεις και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλερ έχει το λόγο. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ε, επιθυμία πως θα ήθελε να έχει ένα μηχανισμό αξιολόγησης για το Σέγγεν και μια τακτή ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό και θα ήθελα να μάθω εάν αυτό υλοποιείται Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε την κυρία Πάικ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέροντα και τα έγγραφα που αφορούν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχω πολλές ερωτήσεις και σχόλια για τις γενικές διατάξεις. Ελπίζω να προλάβω να τις παρουσιάσω. Γενικώ δεν είμαστε κατά Τη σύσταση 2 αντί για 4 ταμεία. Νομίζω ότι έτσι δημιουργείται ένα πιο εύκολο και πιο καλό περιβάλλον, αλλά θέλουμε σαφή κατανομή ανάλογα με τις προτεραιότητες και να ξέρουμε τι περιλαμβάνει κάθε γραμμή. Να μην έχουμε όλα τα κονδύλια για επαναπατρισμό ή για επανεγκατάσταση ή για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι κονδύλια αφιερώνονται σε τι σκοπό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει κάποιο λόγο για το πόσα κονδύλια θα αφιερωθούν σε κάθε προτεραιότητα. Έχω και μια συναφή ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα από την πρόταση, τα κράτη-μέλη θα θεσπίσουν του δικού του στόχου. Υπάρχει ένα διάλογο πολιτική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει γενικού στόχου, αλλά κάθε κράτο είναι αρμόδιο να θεσπίσει του δικού του στόχου ανάλογα με τι ανάγκε του. Έτσι όμω δημιουργούνται περισσότερε αβέβαιε φαίε ζώνε υποβαθμίζεται ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημιουργείται μια τέτοια οριστία, μια φαιά ζώνη και αβέβαιη που απευχόμαστε. Πώς το εξηγείτε. Ποιο θα ορίσει του στόχου, ποιο θα ελέγξει αν υλοποιούνται και με ποια βάση. Επιπλέον, η αναθεώρηση του προπολογισμού που κάπως αργά μας υποβάλλατε, αλλά καλό αργά παραποτέ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κοινοτικά κονδύλια θα αφιερωθούν σε δράσεις που έχουν προστιθέμενη αξία και σε πράξεις που τους άλλους δεν θα μπορούσαν τα κρατη από μόνα τους να χρηματοδοτήσουν. Εδώ θα πρέπει να ε, συμφωνήσουμε ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούμε πράξεις, δράσεις που τους ή άλλως θα κάνουν τα κράτη-μέλη, αλλά εδώ βλέπουμε ότι η Γερμανία χρησιμοποιεί κρατικά, κοινοτικά κονδύλια, συγγνώμη, για νέες ε, θέσεις, ε, για να στελεχώσει νέες θέσεις ε, στο αεροδρόμιο της Νιρεβέρης που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Ή ότι η Ισπανική κυβέρνηση χρησιμοποιηθεί ε, κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση ε, μαθημάτων πρώτη πρώτης ανάγκης. Είναι χρήσιμα με αυτά τα μαθήματα, αλλά δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ούτως ή άλλως έπρεπε η η Ισπανική κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τέτοια μαθήματα, σεμινάρια πρώτης ανάγκης, για παροχή πρώτης ανάγκης. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 60 των Γενικών Διατάξεων, αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει στο 90% αν η δράση αυτή δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί αλλιώς. Αλλά αυτή η διάταξη είναι αντιφατική με την ιδέα ότι μόνο προστιθέμενες, προστιθέμενη αξία και σχετικές δράσεις θα χρηματοδοτήσουμε. Και πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτό το διάλογο πολιτικής που εξήγηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήσασταν πολύ σαφείς για την εξωτερική διάσταση που δεν θα πρέπει να προσανατολίζεται στην ανάπτυξη και ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοχή με τις εξωτερικές δράσεις. Αυτά ήταν όλα πολύ σαφή. Αλλά πώς θα το εφαρμόσετε, αν έχουμε μία ασάφεια ή μία αμφισβήτηση. Ποιος θα αποφασίσει αν πρόκειται για εσωτερικές υποθέσεις ή ανάπτυξη. Πώς θα εξασφαλίσετε εφαρμόγη της συνοχής. Γιατί δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο συμφωνούμε με την ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά χρειαζόμαστε και εξωτερική αξιολόγηση, γιατί τώρα έχουμε εξωτερική αξιολόγηση του προηγούμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά πολύ καθυστερημένα για το τωρινό. Έτσι ουσιαστικά συγκεντρώνουμε τεχνικές παρατηρήσεις και στατιστικές πληροφορίες, αλλά δεν βλέπουμε ε, ποιους στόχους υλοποιούμε. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Παρακολούθησης, πώς θα λειτουργήσει, ποιο θα είναι ακριβώς το έργο της. Και τέλος, αναφέρατε ότι η καταστρατήγηση του κοινωτικού δικαίου θα πρέπει να οδηγήσει σε χρηματοπιστωτικές διορθώσεις μόνο σε περιορισμένες ε, περιπτώσεις. Εγώ φανταζόμουν ότι οποιαδήποτε καταστρατήγηση κοινωτικού δικαίου θα έχει δημοσιονομικές συνέπειες. Κάπου κάτι δεν κατάλαβα φαίνεται. Παρακαλώ, εξηγήστε το. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίρκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στους βασικούς στόχους. Νομίζω ότι αυτά τα μέσα που συζητάμε εδώ μπορούν να είναι μέσα που θα μας διασφαλίσουν, το, που θα μας φέρνουν πιο κοντά στο χώρο ε, ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης γίνεται προσπάθεια για μεγαλύτερη ολοκλήρωση, δηλαδή περισσότερες αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν αποτελεσματικά να ε, υπάρχουν μέτρα για ε, καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα εσωτερικών ε, μετανάστευσης και ασύλου. Επικροτώ την απλοποίηση, αντί για έξι ταμεία να έχουμε δύο. Ε, και με έναν ενιαίο μηχανισμό. Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι έχουμε αύξηση στα ταμεία αυτά. επειδή υπάρχουν νέα κοινοτικά καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να ε, εκπληρώσουμε και στον τομέα ασύλου, μετανάστευση και εσωτερικών. Αν, θέλουμε, αν ζητάμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει ε, να διατεθούν και τα απαραίτητα μέσα. Επίσης, ε, θετικό θεωρώ ότι είναι η αυξημένη ε, ευελιξία. Προβλέπουμε πολιετή προγράμματα, ωστόσο μπορούν να γίνουν ε, προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες. Σημαντικό είναι να υπάρχει πολιτικός διάλογος όχι μόνο στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο ε, μέσο. Ναι, θέλουμε πολιετές ε, πλαίσιο, αλλά με την ε, απαραίτητη ευελιξία, ώστε να μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις όπου είναι απαραίτητο. Θεωρώ επίσης καλό να προβλέπονται περισσότεροι πόροι για την κεντρική διαχείριση. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει από εδώ, ε, στο σημείο αυτό, επίκριση από τα κράτη-μέλη που θα προτιμούσαν κάτι άλλο. Αλλά ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε την ευρωπαϊκή πτυχή. Όταν ε, δούμε πώς είναι οργανωμένη η άμεση βοήθεια, με τη... Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η μέθοδος που έχει επιλεγεί να έχουμε προκαταβολή κατά 4% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, αυξήσουμε την προκαταβολή διότι για μη αποτελεσματικά προγράμματα δεν θα βρεθούν ούτως ή άλλως οι απαραίτητοι πόροι. Ε, νομίζω ότι έτσι έχουμε έναν ε, επιλεκτικό μηχανισμό ώστε να πραγματοποιηθούν τα πραγματικά απαραίτητα προγράμματα, ε, ενώ τα όχι απαραίτητα να μπουν σε δεύτερη μοίρα. Πιστεύω ότι είναι καλό για την άμεση βοήθεια να σκεφτούμε δράσεις ad hoc, οι οποίες θα αποτελούν άμεση αντίδραση εδώ θέλουμε χρηματοδότηση 100%. Θα θέλαμε όμως να προτείνουμε όταν λόγω ε, λήψεων, ε, για παράδειγμα, ε, της για ελλείψεις κατά την συνοριοφύλακη, αν στις περιπτώσεις αυτές ε, καταργηθούν ε, τα μέτρα, τότε θα πρέπει η Κομισιόν να βρίσκει τρόπους ώστε να αποφευθούν οι ελλείψεις αυτές. Το 5% των μέσων προβλέπεται για τεχνική υποστήριξη. Αυτό δεν μπορώ να το ε, εκτιμήσω, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε αν αυτό αρκεί ή όχι. Και ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Πρόκειται για ερώτηση προς την Κομισιόν. Μπορεί να με ενημερώσει, να με διαφωτίσει. Στο σημείο 632 αναφέρεται επιμέρους στόχους του Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Στο σημείο Γ, αναφέρεται η προώθηση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής ε, στα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το δίκαιο μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς, αλλά τι είναι οι αποτελεσματικές στρατηγικές επιστροφής εντός των κρατών μελών. Και στο σημείο Δέλτα μιλάτε για τον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών που θα λάβουν ενίσχυση. Από ό,τι γνωρίζω, έχουμε το Δουβλίνο νομική βάση το οποίο σημαίνει ότι η πρώτη χώρα εισόδου είναι αρμόδια για την διαδικασία ασύλου. Εφόσον έχουμε το Δουβλίνο, γιατί χρειάζεται να γίνει καταμερισμός των ευθυνών. Το Δουβλίνο ορίζει τις ε, ευθύνες. Θα ήθελα παρακαλώ απάντηση στα δύο αυτά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρόν, στη σειρά σας. Θα έλεγα το γεγονό ότι η συμπερίληψη ε, των, ε, των κρατών μελο και ιδιαίτερα του Ηνωμένου Βασιλείου ε, χρηματοδοτεί μερικές φορές εξεγέρσεις σε εξωτερικές χώρες αντί να αφιερώνουμε τα κονδύλια στο εσωτερικό. Ναι, με να, να παρέχουμε καταφύγιο σε ε, πρόσφυγες χωρών ε, που προσπαθούν να ξεφύγουν από την τραγωδία που τους προκάλεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να τους εγκαθιστούμε και μόνοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ε, ξοδεύουμε τα κονδύλια μας για να στεγάζουμε ανθρώπους που προσπαθούν να φύγουν από την ελευθερία και να αποφύγουν τη δημοκρατία. Σε επισφαλείς σχεδίες φτάνουν οι πρόσφυγες αυτοί, να τους δώσουμε σκάφη ασφαλή για να επιστρέψουν στην δημοκρατία και στην ε, νεοπαγή τους ελευθερία. Αυτό δεν είναι που θέλουμε. Αυτό δεν είναι μια, αποτελεσματική πολιτική επαναπατρισμού και επιστροφών. Κυρία Χίρς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γενικά ε, βρίσκω, και... βρίσκω και εγώ θετική τη συγχώνευση των ταμείων. Έτσι έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Ταυτόχρονα μπορώ να συμφωνήσω με τους πράσινους ότι θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα ποσά για τους διάφορους θεματικούς τομείς ώστε να μπορεί ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει βάρος σε κάποιους τομείς ώστε τα κράτη-μέλη ε, να μην ε, μπορούν να αγνοήσουν κάποιους τομείς ή να χρησιμοποιήσουν όλα τα χρήματα για έναν μόνο τομέα. Ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εδώ υπάρχουν ε, διάφορα στοιχεία. Λογικό είναι να ε, δουλεύουμε με εφάπαξ ποσά, τα μικρά προγράμματα μπορούν να λαμβάνουν εφάπαξ ποσά, διότι αλλιώς θα είναι υπερβολικό το άχθος, το γραφειοκρατικό άχθος για τους μικρούς οργανισμούς. Επίσης, τα χρήματα θα πρέπει γρήγορα να φτάνουν στους φορείς εκτέλεσης, διότι είναι γνωστό και από τον κοινωνικό τομέα οι μικρό, μικροί αυτοί φορείς να συναντούν προβλήματα ε, σε περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος ήδη έχει τα λάβει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό θα πρέπει να το φροντίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φατζιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα η συγχώνευση των ταμείων, ωστόσο αυτό δεν ε, θα πρέπει να είναι εις βάρος της αποτελεσματικότητας των ταμείων. Δεν θα πρέπει με τον τρόπο αυτό ε, να περιοριστούν τα διαθέσιμα ποσά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ε, έχω όμως κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά ε, την παρακολούθηση ε, της ε, απελευθέρωσης των πόρων. Σήμερα ήδη αναφέρθηκαν η Λαμπεντούσα και η Σικελία. Επισκέφθηκα ένα από τα κέντρα ασύλου και εκεί είδαμε ότι η Ιταλική κυβέρνηση έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει πολλούς πόρους από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για να βοηθήσει τους πρόσφυγες και λαθρομετανάστευς. Ωστόσο, τα ποσά που τελικά διατίθενται σε κάθε άτομο είναι πενιχρά. Οι ε, πόροι του κέντρου ήταν ανεπαρκείς για την ε, προμήθεια εφημερίδων ε, ή τηλεοράσεων. Κάποιες από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις είχαν υποψίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε την κατάχρηση κατά την κατανομή των ποσών ε, σε διάφορες κυβερνήσεις. Αναρωτιέμαι αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τα ποσά που τελικά ε, διανέμονται σε αυτούς που θα πρέπει, ε, που χρειάζονται τα ποσά αυτά, που θα πρέπει να τα δαπανίσουν για την επιβίωσή τους. Επισκεφτήκαμε και την Αφρική, το Μάλι και άλλες χώρες. Εδώ δαπανώνται χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διατίθενται στις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις όμως είναι διεφθαρμένες και έτσι τα χρήματα δεν φτάνουν σε αυτούς, στους πιο ευάλωτους. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε τα χρήματα να ε, ε, λαμβάνονται από τους πραγματικούς δικαιούχους. Ευχαριστώ. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις η εκπρόσωπος της Κομισιόν, η κυρία ε, Πάικ, ε, παρακαλείται να απαντήσει όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε να έχουμε χρόνο και ε, για το επόμενο θέμα, το οποίο είναι παρόμοιες φύσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ενδεχόμενα να μην απαντηθούν όλες και ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι κάποια θέματα αφορούσαν το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και ο συνάδελφος θα κάνει μια παρατήρηση αργότερα και ενδεχόμενα να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματά σας. Τώρα, για το θέμα της αξιολόγησης, του μηχανισμού αξιολόγησης Schengen του κ. Μίλντερ. Η απάντηση βρίσκεται στο μέσον για το ISF στο άρθρο 13 όπου προβλέπουμε τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή μηχανισμού αν ε, κράτος μέλος ε, πρέπει να αναλάβει δράση σύμφωνα με την αξιολόγηση Schengen υπάρχει ε, πρόνοια για την τροποποίηση του προγράμματος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λαμβάνουν περισσότερα χρήματα επειδή έχουν ελλείψεις υπάρχει το πολιετές πρόγραμμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις. Τώρα σχετικά με τα σχόλια για την κατεπίγουσα βοήθεια, ειδικά μετά όσα συνέβησαν πέρυσι. Λυπάμαι που κάποια κράτη μελεσάνθηκαν εγκαταλελειμμένα. Δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι τέτοιο. με ε, την Ιταλία η οποία επλήγει ιδιαίτερα. Ήμασταν πολύ κοντά στην Ιταλία και προσπαθήσαμε να αποκτήσουν επιπλέον πόρους και για θέματα άμεσης δράσης συζητήσαμε το ζήτημα αυτό. Υπήρχε συνεχής επαφή με τις ιταλικέ αρχέ και το ζήτημα δεν ήταν η έλλειψη κονδυλίων, αλλά έπρεπε να δράσουμε και να δράσει η Ιταλία άμεσα. Καμία χώρα δεν εγκαταλείφθηκε. Υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν φρόντισε από το προηγούμενο του 2011 να χορηγηθούν κονδύλια προκειμένου να δοθεί επιπλέον βοήθεια σε χώρες της Νοτιού Μεσογείου. Υπήρξε ένας, ένα κονδύλι 9 εκατομμύριων ευρώ στην Frontex ε, για περίπτωση που θα χρειαστούν επιπλέον χρήματα ε, στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η κυρία Βίνστρομ αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό ο Γενικός μου Διευθυντής βρίσκεται στην Ιταλία σήμερα. Έχει επαφές με τι αρχές και θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω αν χρειαστεί. Κυρία Κέλλερ έφεξε μια σειρά από θέματα. Νομίζω ότι μιλάτε για την αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος. Λάβατε μια έκθεση, δεν θα σχολιάσω. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει προσθετικότητα στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν έχω λεπτομέρειες για να απαντήσω σε αυτά τα επιμέρους σημεία. Σχετικά τώρα με το πώς διασφαλίζεται ο συντονισμός στην εξωτερική πτυχή. Έχουμε δράσεις σε ευρύτερε χώρες και ενδέχεται κάποια κράτη-μέλη να αναλάβουν δράσεις ε, στη συνεργασία με τα τρίτα χώρα, αλλά η ε, κύρια δράση γίνεται μέσω της άμεσης ε, δράσης της Ένωσης και αυτό πετυχαίνεται με τον κατάλληλο συντονισμό των υπηρεσιών της Κομισιόν και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και υπάρχει συμπληρωματικότητα. Τώρα για τον δύο μέσων. Υπενθυμίζω εδώ τα χρήματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, για τις έκθεση καταστάσεις σε τρίτες χώρες. Παράδειγμα, προβλέπουμε στο άρθρο 9 του κανονισμού πλαισίου ότι συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανώσεις, ε, φορείς ε, των Ηνωμένων Εθνών, την Ερθρό Σταυρό κλπ. Το ότι συνεργαζόμαστε δεν σημαίνει ότι χορηγούμε απαραίτητα και χρήματα σε κάποιε κυβερνήσει τώρα. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλουμε να διασφαλίσουμε ώστε... Τώρα, για τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουμε ξεκινήσει ήδη συζητήσει στην ομάδα ad hoc του Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο η τελική σχέση μπορεί να λειτουργήσει και με ποιο τρόπο ε, η συνεργασία μπορεί να προχωρήσει και ξέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη αισθάνονται ότι ο πολιτικός διάλογος ε, και η συνεργασία ε, μειώνουν κατά την άποψή μας ε, το άχθος, το φόρτο εργασίας και τον οικονομικό βάρος προτιθέμεθα να δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση ειδικά με τον πολιτικό διάλογο, να πούμε ποιος είναι αυτός ο στόχος αυτής της πολιτικής του διαλόγου. Και θα θέλαμε να μάθουμε και το Κοινοβούλιο ποια είναι τα ζητήματα στα οποία επιθυμεί να εστιάσουμε Τώρα για το ζήτημα των στόχων και τους δείκτες ε, ήδη στα επιμέρους μέσα αναφέρουμε παραδείγματα στόχων θα αναπτύξουμε με τα κράτη-μέλη ε, συγκεκριμένους στόχους και δείκτες ε, για κάθε ένα από τα μέσα για το οποίο τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα θέλαν να έχουν ενδείξει. Ε, να ρωτήσω από τον συνάδελφο Στέφανη κάτι να τονίσει κάποιες πτυχές ε, του μηχανισμού ελέγχου και παρακολούθησης. Είναι κάτι που έθιξαν πολλοί βουλευτές ε, συμπεριλαμβανομένου και του εισηγητή. Να δώσω λοιπόν το λόγο στη συνάδελφη Ευχαριστώ Μπελίντα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο το τοπίο για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στην μεικτή, την κοινή διαχείριση. Η πρόταση κανονισμού λαμβάνει υπόψη ένα σημαντικό στοιχείο που είναι η εναρμόνιση με τα υπόλοιπα συστήματα κοινή διαχείρισης. Και φυσικά ε, συνάδει και με την αναθεώρηση του κανονισμού που συνεχίζεται. Έχουμε πλουστεύσει το σύστημα προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμός των αρχών και να, να διευκρινιστούν οι ελεγκτικές αρμοδιότητες. Υπάρχει καλύτερη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί και η ροή των πληρωμών και να φτάνουν πολύ πιο γρήγορα τα χρήματα στους δικαιούχους. Αυτό το στοιχείο ελήφθη καλύτερη υπόψη γιατί το Ταμείο λειτουργεί με ένα μηχανισμό επιστροφής. Δηλαδή θα ε, πρέπει τα διάφορα κονδύλια να καταβάλλονται στους δικαιούχους. Και μετά γίνεται επιστροφή. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε για τις διορθώσεις ε, της οικονομικής στο τέλος, δημοσιονομικές, δεν κατάλαβα και πολύ καλά την ερώτηση. Φυσικά θα γίνουν στο τέλος κάποιες δημοσιονομικές διορθώσεις εφόσον ε, δεν έχουν γίνει σεβαστές οι υποχρεώσεις, η ε, διατάξεις και υπάρχει ένας κίνδυνος η αβεβαιότητα προς την επιλεξιμότητα των κονδυλίων. Πάντως προβλέπεται και τέτοια δημοσιονομική διόρθωση. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ε, να ολοκληρώσει με ένα τελικό σχόλιο ο εισηγητής. Ε, πρόεδρε, σε ό,τι φορά τώρα το ζήτημα θα πρέπει να εμβαθύνω κάποιες ερωτήσεις ε, και τις απαντήσεις φυσικά της Κομισιόν. Είμαι στην διάθεση όλων των συναδέλφων για περαιτέρω συζήτηση επί της εκθέσεως. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Καιρός τώρα για να ολοκληρώσω αυτό το πρώτο σημείο της Μέσης Διατάξεως ε, που αφορά στις παρουσιάσεις ε, για το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Οι εισηγητές ε, έχουν συμφωνήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Ένα εργαστήρι θα οργανωθεί στις αρχές Απριλίου και έκθεση θα συζητηθεί Μάιο ε, Ιούνιο, κατάθεση τροπολογιών τον Ιούλιο και εξέταση των τροπολογιών τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτός είναι προσανατολισμός σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και οι ψηφοφορίες θα γίνουν ε, τον Νοέμβριο. Τώρα φτάσει ό,τι φορά το σημείο 4 για τι γενικέ διατάξει ταμείου για το άσυλο μετανάστευση και μέσω χρηματοδοτική στήριξη. Περνάμε τώρα στα επόμενα σημεία 5, 6 και 7 που είναι τη ιδία φύση. Αφορούν το πολιτέ χρηματοδοτικό πλαίσιο. Περνάμε ω εκ τούτου στο επόμενο σημείο. Η συγητής είναι η κυρία Σιλβίκη Γιώμ για το Ταμείο για το άσυλο και τη μετανάστευση, αλλά πρώτα θα έχουμε μια παρουσίαση από την Κομισιόν, ανταλλαγή απόψε, να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική που εφαρμόσαμε και για το σημείο 4. Θα ακούσουμε λοιπόν από την κυρία Μπελίντα Πάικ της Κομισιόν μια παρουσίαση, μετά την Δανική Προεδρία και μετά την εισηγήτρια. Κυρία Μπελίντα, έχετε το λόγο. Αυτή τη φορά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να κάνει την παρουσίαση για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, πρόταση δηλαδή για την σύσταση ενός τέτοιου Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, έχει στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου περιεκτικού μηχανισμού για να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών, αλλά και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Βέβαια, χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα μέσα και μηχανισμούς και κυρίως τρία από τα ταμεία του Γενικού Προγράμματος για την ελεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά ξεπερνάει και όλα αυτά τα θέματα και προτείνει κάποιες απλουστεύσεις Υπάρχει η απόφαση δηλαδή για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης που καλύπτει από αυτή την πρόταση. Και αν εξετάσουμε την παρούσα κατάσταση με τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πειραματικά σχέδια που εξετάζονται και θα εγκριθούν από την αρμόδια για την προπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης, διαπιστώνουμε ότι η πρόταση αυτή καλύπτει και άλλους τομείς Οπότε η απλοποίηση που γίνεται είναι πολύ πιο φιλόδοξη από την απλή συγχώνευση τριών ταμείων. Επαναλαμβάνω, δεν μιλούμε για μια απλή συγχώνευση των ταμείων, αυτό θα ήταν κάτι γραφειοκρατικό, αλλά θέλουμε με την απλοποίηση αυτή να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ταμείων ε, σε ορισμένους τομείς έχουμε μεγαλύτερη έμφαση της πρότασης, ε, για παράδειγμα στις προτεραιότητες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, όπως είναι τα θέματα επανεγκατάστασης των προσφύγων, η ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ένταξη σε περιφερειακό επίπεδο με κάποιες πολιτικές ένταξεις ή συνδρομή σε περίπτωση που ζητάτε κάτι τέτοιο και γεφύρωση των χασμάτων σε περίπτωση που εντοπίζονται αυτά τα χάσματα, κάτι που δεν επιτρέπει η παρούσα κατάσταση ή δεν το επιτρέπει τουλάχιστον με αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της δράσης μεταξύ των διαφόρων χωρών, της διακριτικής δράσης που αναφέρει η Μπελίντα Πάικ, ή για άλλες δράσεις που αφορούν την νόμιμη μετανάστευση και που αυτή τη στιγμή δεν εμπίπτουν ε, στις επιλέξιμες δράσεις του Ταμείου ε, για τη μετανάστευση. Υπάρχουν πολλά ωφέλη από την συγχώνευση των ταμείων και την απλούστευση της κατάστασης. Έχουμε ένα απλοποιημένο πλαίσιο για τις ομάδες στόχου, γιατί αυτή ήταν μια δυσκολία που αναφέρθηκε πολλές φορές. Για παράδειγμα, στις διάφορες δράσεις ε, ένταξης εστιαζόμαστε σε πρόσφυγες ή υπηκόους τρίτων χωρών που είναι νόμιμοι μετανάστες, αλλά τέτοιες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες από το ίδιο ταμείο. Κάτι που δεν θα ισχύσει πια με το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση που θα καλύπτει και τέτοιες δράσεις έχουμε ένα διευρυμένο ορισμό και της κατεπίγουσας κατάστασης, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι πιο συσταλτική η ερμηνεία που δίνουμε, πιο διασταλτική, συγγνώμη, πιο ευρεία. Ε, ιδιαίτερα για τους υπηκός τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, για τις μικτές ροές και τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης σε τρίτες χώρες. Η πρόταση αυτή προβλέπει και ένα ε, πανευρωπαϊκό, ενωσιακό μάλλον πρόγραμμα ε, πανεγκατάστασης που θα εφαρμοστεί με πολύ δυναμική διαδικασία και με προτεραιότητες που θα θεσπίζονται αναδιετία με βάση έναν μηχανισμό που είναι παρόμοιος με το μηχανισμό που ευελπιστούμε ότι θα οριστικοποιηθεί ε, το μήνα αυτό για το νέο πρόγραμμα επανεγκατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα θα γίνει ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τέλη του μήνα, όπως σας είπα. Ε, η πρόταση περιλαμβάνει και την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, όπως προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου του 2008, εμπίπτει και αυτό το ταμείο στο ταμείο για το άσυλο, και αυτό το δίκτυο στο ταμείο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Και το δίκτυο αυτό είναι ανοιχτό προς την κοινωνία των πολιτών, τους πανεπιστημιακούς κύκλους και άλλους φορείς που σχετίζονται με την εφαρμογή πολιτικών σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Αναφέρθηκε επίσης ότι το Ταμείο θα έχει και μία συνιστόσα διακρατικών δράσεων. Αναφέρθηκε αυτό και στο οριζόντιο οργά μηχανισμό, δεν θα το αναπτύξω περαιτέρω. Τώρα για το ποιες δραστηριότητες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Είναι πολλές και διάφορες. Πάντως υπάρχουν κάποιοι τομείς που είναι υποχρεωτικοί για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή δράσεων στο άσυλο και στην εφαρμογή του κοινού προγράμματος συστήματος ασύλου σε θέματα εφαρμογή στρατηγικών ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ε, για τις επαναπατρισμούς, για τους ε, οικειοθελείς επαναπατρισμούς και στα πλαίσια της ε, αλληλεγγύης και της ε, κατανομής των ε, υποχρεώσεων με τα θέματα της μετεγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά τα ποσά, το συνολικό ποσό είναι λίγο χαμηλότερο από 4 δισεκατομμύρια, δηλαδή 3 εκατομμύρια 3 δισεκατομμύρια 900 εκατομμύρια και 3,2 δισεκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν προγράμματα των κρατών μελών. Δηλαδή το 84% του συνολικού κονδυλίου θα χρηματοδοτήσει προγράμματα των κρατών μελών και το υπόλοιπο 16% θα το χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια μιας ε, κεντρικής διαχείρισης για διάφορες δράσεις όπως σας ανέφερα ε, ε, συνδρομή ανάγκη, εξωτερική δράση και δίκτυο, ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά τα ποσά που χορηγούνται στα κράτη-μέλη, 74% θα χορηγηθεί ως βασικό ποσό στα κράτη-μέλη στις αρχές της δημοσιονομικής ε, περίοδου που καλύπτει το πρόγραμμα και το 26% θα εξαρτηθεί από την προθυμία των κρατών μελών να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ε, και δράσεις που έχουν προτεραιότητα στους μηχανισμούς αυτούς, ιδιαίτερα θέματα επανεγκατάστασης ε, ή επανατοποθέτησης και συγκεκριμένες δράσεις, 21% των κονδυλίων που αφιερώνονται στα κράτη-μέλη και το υπόλοιπο 5% ε, το αφήνουμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτό είναι σημαντικό για τη δεδομένη τη παρούσα κατάσταση, όπου πολλέ οργανώσει έχουν προβλήματα ω προς τι πληρωμές και τι διαδικασίε πληρωμών, γιατί τα ετήσια προγράμματα στα βασικά ταμεία δημιουργούν μια κατάσταση αναμονής για τους δικαιούχου που δεν ε, μπορούν να λάβουν τα κονδύλια μέχρι ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για να λάβουν τις τελικέ πληρωμές από τις αρμόδιες αρχές. Με τη νέα πρόταση η κατάσταση αλλάζει. Γιατί τώρα πια τα κράτη-μέλη θα μπορούν να στέλνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο αίτημα πληρωμής και μπορούν αυτή η αίτηση πληρωμής να περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληρωμή καταβάλλεται σε εφαρμοστικούς οργανισμούς. Προχρηματοδότηση, ενδιάμεσες πληρωμές και τελικές πληρωμές. Δεν χρειάζεται να περιμένουν τις τελικές πληρωμές οι δικαιούχοι. Θα ήθελα να απαντήσω τώρα σε μία ερώτηση που τέθηκε στην προηγούμενη έκθεση. Είπαμε ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο, προσημειωμένο ποσό για, για τον κάθε τομέα πολιτικής. Αυτή είναι εσκεμμένη επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφύγει κάποιες διοικητικές περιπλοκές στη διαχείριση του Ταμείου. Τέτοιες περιπλοκές φυσικά είναι περιττές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αμελήσουμε κάποιες πολιτικές στην εφαρμογή των κονδυλίων. Υπάρχουν κάποιες, κάποιοι τομείς που είναι οριοθετημένοι. Υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά προσδιορισμένα για την επανατοποθέτηση και τη μετεγκατάσταση, καθώς και για συγκεκριμένες δράσεις. Αυτά τα ποσά θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον τα κράτη-μέλη δεχτούν να συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Και όπως είπα, υπάρχουν και κάποιοι τομείς που είναι υποχρεωτικοί και άλλοι που είναι προαιρετικοί. Το άσυλο είναι ένας από αυτούς, τους προαιρετικούς. Σε ό,τι αφορά τα ποσά της κάθε πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των συγκεκριμένων αναγκών κάθε χώρας, γιατί σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και το μέγεθος των μεταναστευτικών ορών υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και θα θέλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγουμε έναν άκαμπτο κανόνα που θα ισχύει για όλους άσχετα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους. Το άρθρο 20 λοιπόν καθιστά υποχρεωτικές μόνο ορισμένες από τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ <clears throat> για την ενδελεχή παρουσίαση. Περνάμε τώρα στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, κυρία Κίτρον Μέλλα. Ευχαριστώ. Η Προεδρία εν συντομία μπορεί να σχολιάσει σήμερα σχετικά με αυτή την πρόταση για το Ταμείο Περιασύλου και Μετανάστευση. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στον αρμόδιο στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου είχαμε την δυνατότητα να ζητήσουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες, θέσαμε ερωτήσεις για διευκρινήσεις κλπ. Περάσαμε στην πρώτη ανάγνωση τον Φεβρουάριο και θα συνεχίσει την προσεχή εβδομάδα. Να πω ότι τα κράτη-μέλη γενικά ε, καλοδέχθηκαν ε, την πρόταση της Κομισιόν και την ε, δυνατότητα συγχώνευσης των τριών ταμείων σε ένα, κάτι το οποίο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελεξία στην διαχείριση των ταμείων τα κράτη-μέλη ε, εξετάζουν το πεδίο εφαρμογή ε, της ε, πρότασης και τις επιπτώσεις που θα έχει σε διοικητικό επίπεδο και την αλλά και άλλες λεπτομέρειες της νέας πρότασης. Η συζήτηση λοιπόν που σας είπα ξεκίνησε το Φεβρουάριο στο Συμβούλιο, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα, αλλά η Προεδρία προσβλέπει σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο επί του θέματος και φυσικά Είμαστε στην ε, διάθεση των ε, εισηγητών, όπου αυτοί το κρίνουν απαραίτητο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και την Προεδρία. Ξεκινάμε τώρα με την εισηγήτρια, κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικά επιπλέον σχόλια μετά από την παρουσίαση της έκθεσης, η οποία ήταν πληρέστατη, δεν θα επανέλθω. Να πω όμως ε, ότι προτείνονται κάποιες ε, βελτιώσεις που πάνε προς την κατεύθυνση. Καταγράφω την ε, δήλωση για, μια πολυε... για έναν πολυετή προγραμματισμό. Νομίζω ότι είναι ε, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια, ειδικά σε όσους επιθυμούν να μην βρίσκονται σε επισφαλή θέση κατά την καθημερινή τους δραστηριότητα τη συμπερίληψη του υποχρεωτικού κριτηρίου, ιδιαίτερα αναφορικά με το θέμα των επιστροφών, με μία έμφαση στον, στον όρο εθελούσια επιστροφή. Να πω επίσης για την προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και στην ε, ένταξη, διότι αυτό το συζήτησαμε με τη διάρκεια της προηγούμενης έκθεσης, αναφορά σε έκτακτες καρδίγους καταστάσεις ε, που προσδιορίζονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αναφορά στις κατεπίγουσες καταστάσεις και τον τρόπο της ε, καλύτερης δυνατής ε, ανταπόκρισης. θα είναι τα σημεία που θα ήθελα να τονίζω. Έχω κάποια ερωτηματικά παρατηρήσεις που θα σας αναφέρω και που θα απαντήσουν ε, στο οποίο θα απαντήσει και η Κομισιόν όπως έπραξε τις προηγούμενες συνεδριάσεις αλλά και θα ακούσουμε και τις θέσεις των ε, σκιωδών εισηγητών τώρα το θέμα του ασύλου η Κομισιόν τόνισε το ζήτημα της επανεκατάστασης ε, για, και για να, δω, για να χορηγήσει στήριξη στα κατημέρια. Ξέρουμε ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη ε, εργάζονται, εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου και θα πρέπει να μειώσουν αυτόν τον φόρτο εργασίας αλλά η εξέταση των πολλαπλών αυτών αιτήσεων ασύλου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα μια ερώτηση για το ζήτημα της ένταξης, διότι κατάλαβα ότι ένας από τους υποχρεωτικούς στόχους, όπως ανέφερε η Κομισιόν, ήταν να προβλέπεται η στήριξη των περιφερειακών πολιτικών ε, ένταξης και ε, ενσωμάτωσης με τις περιφερειακές αρχές ε, και φορείς και αν έτσι έχουν τα πράγματα θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδέσουμε αυτούς τους τοπικούς φορείς στον διαδικασία προγραμματισμού. Θεωρώ πως η εμπειρία τους ε, θα έχει πολλά να προσφέρει. Το, το Ταμείο ε, κεντρώνεται στο θέμα της ε, αλληλεγγύης, ε, τονίστηκε, αλλά δεν υπάρχει μνήμα του άρθρου 80 της συνθήκης ως νομική βάση και θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν ε, δράξαμε την ευκαιρία να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση ε, και άλλα δύο σημεία εντάχει. Όπως είπε ο κύριος Σινιώρε προλίγου, η Γενική Διεύθυνση ε, εξετάζει το θέμα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων και με κάνει αυτό να επανέλθω σε ένα ζήτημα για ενδεχόμενη σύγχυση με άλλες μορφές ε, δράσης, ε, την ανθρωπιστική κλπ. Θα ήθελα λοιπόν τα πράγματα να γίνουν ξεκάθαρα μετά από τις συζητήσεις μας. Και τέλος, ε, Ο κ. Σινιόρ μίλησε για ισορροπία, για μην ε, προηγούμενη δέσμευση των ε, κονδυλίων. Καταλαβαίνω αυτή την διάθεση ε, ευελιξίας, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ότι ορισμένες πτυχές και ειδικά η πτυχή ένταξης δεν μπορεί να περάσουν στην τελευταία θέση είναι θέμα στο οποίο είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Και τώρα περνάμε στις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων. Κοιτάξτε, έχουμε καθυστερήσει ήδη 20 λεπτά. Σύντομη παρακαλώ να είσαστε. Κυρία Βέλστρομ. Η κυρία Βίκστρομ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις πληροφορίες που μας έδωσε για το νέο αυτό Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από την Κομισιόν σχετικά με το αν προβλέπονται διατάξεις ε, για να υπάρξει σχετικά με το άρθρο 13 ε, στον κανονισμό του Βλήνο 2 ε, για περιπτώσεις ε, άμεσης παρέμβασης στο άρθρο 6 της πρότασης για τη δημιουργία του Ταμείου για, το άσυλο και τη μετανάστευση είδα την εξής διατύπωση. Τα Η δυνατότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές ασύλου τους η ερώτησή μου είναι, αυτό αναφέρεται σε ανάπτυξη νέων πολιτικών, όπως είναι η δημιουργία ενός ε, μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης ε, στον κανονισμό Δουβλίνο 2 ή ε, αναφέρεται σε κάτι άλλο. Η Κομισιόν έχει προβλέψει γραμμή του προϋπολογισμού για αυτόν τον νέο μηχανισμό. Ιδιαίτερα δεδομένου του γεγονότος ότι θα αυξηθεί το άρθρος εργασίας του ΙΑΣΟ και μάλιστα ριζικά. Αυτή είναι η σύντομη ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αρκετά θέματα ήδη αναφέρθηκαν. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Στο άρθρο 19 του οριζοντίου κανονισμού ε, αναφέρεται η απαγόρευση ε, οικοπαίδων. Στο άρθρο 5, παράγραφος 2α, υπάρχει ε, η προϋπόθεση ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εστέγασης. Υπάρχει νομικός λόγος ε, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται η απαγόρευση η αγοράς οικοπαίδων. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει νομικός ε, λόγος που, είχε που έχει αφαιρεθεί ε, η ε, απαγόρευση της αγοράς σκοπέδων από τον βασικό κανονισμό. Επίσης, δεν συζητάμε εδώ την κράτηση σε φυλακές. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια να πρέπει υπό κάποιες προϋποθέσεις ε, να στεγαστούν σε νέα κτίρια. Ε, δεν έχω καταλάβει, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη συνέπεια ανάμεσα στα δύο αυτά κείμενα. Και επίσης ερώτηση στο άρθρο 3, εδώ αναφέρονται κάποιοι στόχοι. Στο 2 δέλτα αναφέρεται η αλληλεγγύη και ο καταμερισμός ε, της ευθύνης. Αυτό αναφέρεται ε, στην εθελοντική ανταλλαγή ε, ετούντων ασύλου. Αγγίζουμε εδώ ελαφρά τον Τουβλίνο 2. Τα κράτη-μέλη μπορούν εθελοντικά να κάνουν κάτι τέτοιο. Πώς πρέπει να το καταλάβουμε το σημείο αυτό. Ωραία. Η κυρία Ολμαϊρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ε, χαίρομαι ότι έχουμε εδώ πιο σαφή ε, ορισμό του Ταμείου για το άσυλο και τη μετανάστευση. Υπάρχουν κάποια δύσκολα ερωτήματα εντός των κρατών μελών σε σχέση με το πακέτο ασύλου. Ε, διότι ε, συνεπάγεται αυτό και επιπλέον χρηματοδότηση. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Καταρχήν θα πρέπει να συζητήσουμε εντατικά πώς ε, θα γίνει η κατανομή, με ποια κριτήρια θα γίνει η κατανομή ε, οικονομικών μέσων στα κράτη-μέλη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό απόλυτα. Ε, δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι παρόμοιο με αυτό που είπε η συνάδελφος Χίρς. Και εγώ πρόσεξα κάποια σημεία όπου ο κανονισμός αυτός φαίνεται να αντίκειται με τις υπόλοιπες διατάξεις. Ε, θα θέλαμε μία ε, συνεπή νομοθεσία και να μην έχουμε εδώ συγκρούσεις, ώστε και κατά την εφαρμογή ε, στα κράτη-μέλη να ξανασυναντάμε δυσκολίες να αναφερθώ στους συγγενείς ή το θέμα που ανέφερε η κυρία Χίρς. Το ότι συμπεριλαμβάνονται εδώ και οι αιτούντες άσυλο. Ε, ε, όταν μιλάμε για παράδειγμα για την θελοντική ανταλλαγή. Θα πρέπει για να είναι αποτελεσματικό το μέσο να υπάρχει συνέπεια και σαφήνεια εντός του πακέτου Πάντως προσβλέπω στην καλή συζήτηση και ελπίζω και στην γρήγορη εφαρμογή του κειμένου. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, σήμερα θα μιλήσω την Πορτογαλική. Πρόκειται για μια ερώτηση γενικότερης φύσης. Ε, μιλάμε για ταμείο για το άσυλο και θα ήθελα να ασχοληθώ με το ζήτημα επανεγκατάστασης ε, των ετούνων άσυλο. Καταρχήν, ε, μια πρώτη γενική ερώτηση, κατά την άποψή μου, κατά τις ανησυχίες της Κομισιόν που θέλει να έχει ένα πιο ευέλικτο ταμείο και ένα ταμείο καλύτερα πρικοδοτημένο αλλά χρειάζεται και ένας ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος σχετικά με το τι γίνεται με το λόγο ταμείο και ποιε είναι οι προτεραιότητε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί στο ζήτημα του καθορισμού των προτεραιοτήτων. Διαφορετικά, ένα ικανό κομμάτι των κονδυλίων θα πηγαίνει στις επιστροφές. Ε, ε, χρειάζεται λοιπόν το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί περισσότερο με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καλά στοχευμένη πολιτική και να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ταμείο. Και κάτι ακόμα, ε, ε, μη κυβερνητικέ μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, θα μπορούσαν και αυτές ε, να λαμβάνουν κάποια κονδύλια, όχι μόνο οι διεθνείς οργανισμοί και αυτό είναι κάτι το οποίο υπόθηκε από την κυρία Κιγιόμ και κρίμα που το άρθρο λοιπόν 80 για την ε, ενδοενωσιακή αλληλεγγύη δεν αναφέρεται διότι αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς επιθυμούμε να ε, πετύχουμε μέσω της χρήσης ε, του Ταμείου. Τώρα, σε ό,τι φορά την ένταξη, όπως αυτή υπήρχε προηγούμενα θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρξει μια μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Ορισμένα κράτη χρησιμοποιούν το Ταμείο Ένταξης για μετανάστες που έχουν ενταχθεί, έχουν νομιμοποιηθεί, έχουν περάσει και το δοκιμασία ε, ε, γλωσσικής επάρκειας ε, κλπ. Πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο τους μετανάστες που βρίσκονται στην πρώτη φάση της ένταξης ε, από την Χαίρομαι που ακούω ότι έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκατάστασης των μεταναστών και θα ήθελα να γνωρίζω αν πέραν των προϋποθέσεων αυτών θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε και κονδύλια για άλλες δραστηριότητες ε, όπως συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους μετανάστες ε, και για, ακόμα για τις υποδομές που απαιτούνται για τα ε, υφιστάμενα κέντρα. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς θα γίνει η διαμόρφωση των κονδυλίων αυτών, πώς θα χορηγηθούν και που αφορούν επίσης και την ε, επίπεδο προετοιμασίας ε, των ε, κρατών. Υπήρχαν χώρες που δεν είχαν την απαραίτητη υποδομή και τους χορηγούμε κονδύλια για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πού ακριβώς πηγαίνουν τα χρήματα. Αλλά εδώ η Κομισιόν κάνει μια πρόταση εντελώς διαφορετική. 6.000 για κάθε είδος ε, εγκατάστασης ε, και 10.000 ε, για κάποιους γεωγραφικούς προσανατολισμούς κλπ. Νομίζουμε ότι είναι κάπως ακραία τα όσα αναφέρονται στην περίπτωση αυτή. Το πρόγραμμα επανεγκατάσταση ξέρουμε ότι είναι από τις φάσεις που είναι πλέον δαπανηρές. Εντάξει, δεν μιλάμε για την Δανία, παραδείγματος χάρη, η οποία έχει ε, πολλά κράτη εμπειρία σε αυτό το ζήτημα. Για μένα λοιπόν αυτή η κατανομή δεν είναι σωστή, είναι κατακαιρματισμένη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την, τον περιφερειακό χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι η Κομισιόν θέλει να περάσει από κατεξουδότηση πράξης, αλλά Ξέρουμε ότι αυτό οδήγησε σε διαφωνίες. Για ένα χρόνο, καθυστερήσαμε λόγω των διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Χρειάζεται λοιπόν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν για τις ε, περιφέρειες, περιοχές που έχουν προτεραιότητα. και μπορεί να υπάρξουν τέτοιες ε, περιοχές ε, σε επίγουσες καταστάσεις, αλλά αυτό όχι μέσω κατεξιότητας πράξεων. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν ε, διαφορετικές δυσκολίε. Κάθε φορά που έχουμε ε, περιπτώσει εκτάκτου ανάγκης, προβλέπεται μια κάλυψη διετής. Εδώ καλό θα ήταν να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κατεξουδότηση πράξη να ορίζει, να χαρακτηρίζει μια τέτοια περίπτωση τη εκτάκτου ανάγκη και μετά να δίνει μια προθεσμία στο Κοινοβούλιο για να αποφαίνεται. Τέλο, το σημείο 5 ε, του παραρτήματος για τις ε, προτεραιότητες, τις δράσεις κατά προτεραιότητα, σε ό,τι αφορά τους ιρακινού πρόσφυγες στη Συρία, Λίβανο και Ορδανία. Παρακαλώ προσέξτε, ένα μεγάλο τμήμα των προσφύγων που προέρχεται από το Ιράκ και βρίσκονται στις χώρες αυτές δεν είναι Ιρακινοί πρόσφυγες, είναι Παλαιστίνοι πρόσφυγες που διέμεναν στο Ιράκ. Να λέμε δηλαδή πρόσφυγες ε, που έρχονται από το Ιράκ, όχι Ιρακινοί πρόσφυγες. Γιατί δεν είναι κατά ανάγκη ε, πρόσφυγες με Ιρακινή υπηκότητα. Επίσης, οι επιβιώσαντες ε, οι θύματα βιοπραγιών και βασανιστήριων δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, γιατί το κατά των δράσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει δύο αντιφατικές στάσεις για την μετανάστευση. Όταν μιλάει στην κοινή γνώμη, λέει ενίσχυση τη διαχείριση του συνόρων. Υπάρχει στην έκθεση αυτή. Και μια βιώσιμη και αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Και ταυτόχρονα ε, υιοθετεί πολιτικές που αντιβαίνουν σε αυτούς τους στόχους που προανέφερε και στις προηγούμενες πολιτικές. Όταν ένας λαθρομετανάστης φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να επαναπατριστεί. Όταν χώρες όπως η Ιταλία προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, ε, συγκέντρωσαν την οργή και την μορφή των υπόλοιπων χωρών. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια νέα απάντηση για το άσυλο, άσχετα με το αν είναι έγκυρη αιτήση ή όχι. Σε ό,τι αφορά την αρχή της μη ε, αποπομπής, της μη απέλαση ε, η επιστροφής, φαίνεται ότι περιλαμβάνεται στη συνθήκη για την εφαρμογή ε, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς, και για την ε, συνθήκη και για την Ένωση, γιατί είναι μια ε, παράλογη αρχή που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να αποπευθεί να επιστραφεί σε επικίνδυνη χώρα. Ενώ υπάρχουν πολλές επικίνδυνες χώρες και αν δεν μπορούμε να επαναπατρίσουμε ένα λαθρομετανάστη σε μια επικίνδυνη ε, χώρα, πώς θα αφήσουμε τους υπόλοιπους πληθυσμούς σε αυτές τις επικίνδυνες χώρες. Να ανοίξουμε τις πύλες μας στο, στο σύνολο του πληθυσμού του Πακιστάν, του Αφγανιστάν ή καταπιεστικών καθεστώτων όπως η Κίνα ε, και να τους φέρουμε όλους στην Ευρώπη μέχρι του βουλιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το βάρος αυτών των πληθυσμών. Αλλά συνεχίζεται αυτή η αρχή λέγοντας ότι απαγορεύεται η επιστροφή, ο παραπατρισμός ακόμη και σε ασφαλείς χώρες. Τότε γιατί δεν επιστρέψαμε Λίβιους και την στα, στους νεοπαγείς παραδείσους ε, και τα λιμάνια δημοκρατίας και ελευθερίας, μια και χώρες αυτές, η Λιβύη και την Ισία, είναι πια ασφαλείς χώρες. Ευχαριστώ. Κύριος Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο παράρτημα της έκθεσης αυτής προβλέπεται μία κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών. Τα κριτήρια αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία ε, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είναι το άσυλο ή όταν ε, απειλείται επιστροφή και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι το κράτος λαμβάνει κονδύλια ανάλογα με τον αριθμό των ε, ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τη γεωγραφική θέση, εξαρτάται και από την κατάσταση της ασφάλειας των συνόρων στις χώρες αυτές. Ερωτώ λοιπόν, πώς θα πρέπει να προβλέψουμε μια αιρεσιμότητα για την κατανομή αυτών των κονδυλίων, ανάλογα με το πόσο βελτιώνεται η ασφάλεια της διαχείρισης των συνόρων και τη σταδιακή μείωση των ατόμων με προβλήματα ασύλου, μετανάστευση και το καθεξής. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν ε, ερωτήθηκε επανειλημμένα για κάποια ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν από την Κομισιόν να απαντήσει. Ehm, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τα περισσότερα σχόλια, μάλλον δεν θα τα καταφέρω να καλύψω όλα τα σχόλια. Η συγκήτρια κυρία Γκυγιόμ είπε ότι υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε τις ε, τρέχουσες δράσεις, όπως αυτές που καλύπτονται από το Ταμείο Προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και θα συνεχίσουμε τις δράσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα περιμένει περισσότερα κονδύλια για τις τρέχουσες ε, δραστηριότητες ε, του Ταμείου Προσφύγων, όπως ε, προβλέπει και το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό και τα ποσά για την επανεκατάσταση και επανατοποθέτηση έχουν προσημειωθεί σε ξεχωριστή γραμμή. Σε ό,τι αφορά την διάσταση της ένταξης, θα πρέπει να αναμειγνύονται οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς το συντομότερο δυνατό στη διαδικασία γιατί ε, συμμετέχουν και μπορούν καλύτερα να εξασφαλίσουν εφαρμογή. Λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο προγραμματισμού και στο άρθρο 9 προβλέπεται μια διαδικασία με ανάμειξη των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων που θεωρείται απαραίτητη. Αναφέρθηκε και το άρθρο 8 ως πιθανή νομική βάση για τα μέσα αυτά. Θα ήθελα να πω ότι το άρθρο 18, συγγνώμη, αναφέρθηκε το άρθρο 18 και το επεξηγητικό με ιδιαίτερη σελίδα 5. Αναφέρεται λοιπόν το άρθρο 18 πιθανή νομική βάση για να υπενθυμίσουμε ότι η πολιτική αυτή και η εφαρμογή τους θα διέπεται από την αρχή της ε, αλληλεγγύης και του καταμερισμού των ευθυνών, αλλά και του καταμερισμού των δημοσιονομικών επιπτώσεων μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητο να περιλάβουμε και το άρθρο 80 στη νομική βάση. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι νομικές βάσεις των διαφόρων πολιτικών θεωρούνται επαρκείς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί πως το άρθρο 80 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως νομική βάση. Όπως προβλέπει μια πρόσφατη δήλωση μετά από τις εξελίξεις για το πρόγραμμα ε, επανεγκατάστασης. Πάντως, σε νομική βάση για τις διάφορες πολιτικές ε, ε περιλήφθηκαν ως κατάλληλες νομικές βάσεις για την εξωτερική διάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε επανάληψη και επικάλυψη δράσεων άλλων φορέων στα πλαίσια του κεφαλαίου 4 του προϋπολογισμού αλλά θέλουμε στην εργαλειοθήκη μας να, περιορίσουμε, να, να, να περιλάβουμε ένα περιορισμένο αριθμό πόρων, κονδυλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να συμπληρώσουν την εφαρμογή δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχει ανάγκη ε, για προσθήκη κάποιων διακρατικών μέσων. Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα με τις δράσεις ε, του κεφαλαίου 4. Η κυρία Βουίκστρομ, ρώτησε το κατά πόσο τα μέσα αυτά θα δημιουργήσουν ένα μηχανισμό αντίστοιχο με αυτόν της πρότασης για τον κανονισμό Δουβλίνο 2. Αυτό ισχύει και για άλλα σημεία που αναφέρθηκαν. Τα μέσα αυτά, τα εργαλεία αυτά θα δημιουργήσουν ένα ελαστικό πλαίσιο για την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης και θα συμπληρώσει κάποιες εξελίξεις στις πολιτικές ε, για την περίοδο 2014 έως 2020, ίσως και μέχρι, μέχρι και το 2022 που είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής του Ταμείου θέτοντας στη διάθεση των ενδιαφερομένων τα κατάλληλα νομικά κονδύλια για να υλοποιηθούν αυτές οι εξελίξεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση δράσεων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων, αξιολόγηση, ιδιαίτερα για τους ε, ετούντες άσυλο, αλλά όχι μόνο για αυτούς. Και φυσικά κάτι τέτοιο θα είναι χρήσιμο όταν εφαρμοστεί ο κανονισμός, γιατί θα θέλαμε το Ταμείο να στηρίζει τις πληροφορίες ε, των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες. Πάντως υπάρχουν τα μέσα και οι μηχανισμοί, υπάρχουν τα εργαλεία για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν στην ΑΖΟ σωστές, ακριβείς πληροφορίες στο μέτρο που αυτές απαιτούνται για την εφαρμογή του μηχανισμού. Η κυρία Ολμάγερ είπε ότι ο ορισμός θα πρέπει να συνάδει με τους ορισμούς της οδηγίας, φυσικά. Και αυτό είναι το ζητούμενο και από εμά. Θα πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι πολλές φορές ο ορισμός της οδηγίας αφήνει κάποιο περιθώριο λιγμών στα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα για την ρήτρα όταν αναφέρεται το, το δύναται. Ε, όταν λέμε δύναται, αφήνουμε ένα περιθώριο λιγμό στα κρατημέλη και τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να προσαρμόζονται στις διάφορες καταστάσεις με ελαστικότητα για να έχουμε αποτελεσματική εφαρμογή. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή της εστίασης των μέτρων ένταξης. Για τις ορισμένες χώρες οι αιτούντες άσυλο περιλαμβάνονται στα μέτρα ένταξης και σε άλλα όχι. Θέλουμε λοιπόν να αφήσουμε περιθώριο λιγμό στα κρατη και να συνεχίσουν πολιτικές και πρακτικές που ευθυγραμμίζονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Πάντως, οι ορισμοί θα πρέπει να είναι αρκετά ελαστικοί, ακριβώς για να καλύπτουν περισσότερες καταστάσεις σε περισσότερα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ταβάρες αναφέρθηκε στο θέμα της επανεγκατάστασης. Όντως έχουμε μια σημαντική εργαλειοθήκη σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις της επανεγκατάστασης των κρατών μελών, γιατί καλύπτονται όχι μόνο οι δραστηριότητες επανεγκατάστασης που χρηματοδοτούνται από το, άρθρο, από το Ταμείο συγγνώμη, και το άρθρο 7 προβλέπει ότι το, όταν το κρατός είναι έτοιμο να αναλάβει επιχειρήσεις ε, επανεγκατάστασης λαμβάνει ένα καταποκοπή ποσό που δίνει έναυσμα και επιβραβεύει ουσιαστικά στα κράτη-μέλη που καταφέρουν να επανεγκαταστήσουν όλο και περισσότερους πρόσφυγες. Και υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα ειδικά εργαλεία που περιλαμβάνει η πρόταση. Το γεγονός, ας πούμε, ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να λάβει συμπληρωματική χρηματοδότηση για να ε, συστήσει κάποια κέντρα διαμετακόμισης. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το εργαλείο είναι αρκετά εκλεπτισμένο και εξυπηρετεί το σκοπό των φιλόδοξων προγραμμάτων επανεγκατάστασης. Ό,τι αφορά την κατεξουσιοδότηση, τις κατεξουσιοδότηση πράξης που τις χρησιμοποιούμε για την αναδιατία θέσπιση των προτεραιοτήτων επανεγκατάστασης. Η συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο για τα θέματα αυτά είναι αρκετά επίμαχη Φάνηκε αυτό το 2009 όταν επισημάνθηκε και εντοπίστηκε αυτή η ανάγκη. Ελπίζουμε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, συμφωνήσουμε, να συμφωνήσουν για να έχουμε μια δυναμική εξέλιξη αυτών των προτεραιότητων. Έχουμε και τώρα κάποιες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ή κατεπίγουσες. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε να προσθέσουμε στον κατάλογο του άρθρου για τα καταποκοπή ποσά, 17 παράγραφος 4, προβλέπεται και η δυνατότητα συμπληρωματικών κονδυλίων για επανεγκατάσταση ε, ή της ε, κατεπίγουσης επανεγκαταστάσεις και τους χρήζοντες βοήθεια. Έτσι καλύπτουμε τις κατεπίγουσες περιπτώσεις, κατεπίγουσες επανεγκαταστάσεις. Τέθηκε και μία ερώτηση για τα θύματα βασανιστήριων και κατά πόσο καλύπτουν και αυτά τα θύματα. Φυσικά τα βασανιστήρια δεν αναφέρονται ρητά, αλλά η πρόταση μιλάει για ευάλωτες ομάδες και ευάλωτες καταστάσεις, ανήλικες, ε, θύματα σωματεμπορίου, γενικώ ανήλικους σε δύσκολες καταστάσεις και προβλέπει διάφορα τμήματα χρηματοδότησης, ε, άσυλο μετανάστευση, επιστροφές, επαναπατρισμό και επανεγκατάσταση. Σε ό,τι αφορά τα ποσά που ρώτησε ο κύριος Μαρινέσκου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να αποφύγει μια ε, επαχθή δημοσιονομική διαδικασία με, την κατέτος, με τον κατέτος προσδιορισμό των κονδυλίων με βάση τα πρόσφατα στοιχεία των κρατών μελών. Γι' αυτό προτείναμε τα βασικά ποσά ε, που δίνονται στα κράτη-μέλη να στηρίζονται σε πρόσφατες στάσεις των μεταναστευτικών ροών. Για παράδειγμα, αριθμό, ε, τον αριθμό των άσυλων, αριθμό νομίμων μεταναστών, ε, αριθμό δυνάμει, δυνητικών μεταναστών, λαθρομεταναστών και ούτω καθεξής. Θέλουμε πολιτι... πολιετή προγράμματα που θα είναι αντίστοιχα με τις μεταναστευτικές ροές των κρατών μελών. Βέβαια, αυτό δεν θα είναι το μόνο εργαλείο. Θα έχουμε και ενδιάμεση αναθεώρηση. Η δυνατότητα ενεργοποίησης της κατεπίγουσας συνδρομής. Έχουμε και τους οργανισμούς Frontex και EASO που επίσης θα μπορούσε να συμβάλλουν σε περίπτωση ιδιαίτερης πίεσης. Και σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα, δεν περιλήφθηκε στο θέμα των ε, ροών ασύλου και μετανάστευσης, αλλά προσφέρει ένα ελαστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις διάφορες συνιστώσεις τους. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Σωτερικής Ασφάλειας και τη συνιστόσα των συνόρων, Εκεί στην παρουσίαση θα σας εξηγήσουμε πώς συνδυάζεται αυτό το θέμα με τη σωστή εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν και τη διαχείριση στο χώρο Σέγγεν. Αυτά και επειδή με πιέζει ο χρόνος λέω να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ για να κλείσουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε την εισηγήτριά μας τη Μαντάμ Κιγιόν. Θέλετε να δευτερολογήσετε, όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Τότε όπως κάναμε και με το προηγούμενο σημείο, θα κάνουμε το ίδιο και για τα σημεία 6 και 7, τα οποία είναι παρόμοια φύση. Στις τέσσερις προτάσεις ε, τις οποίες συζητάμε σήμερα, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στον τομέα θεμάτων δικαιοσύνης και εσωτερικών. Οι εισηγητές συμφώνησαν χρονοδιάγραμμα. Ε, εργαστήριο τέλη ε, Απριλίου, σχέδιο έκθεση Μάιο-Ιούνιο, ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών Ιούλιο, εξέταση τροπολογιών Σεπτέμβριο το αργότερο, τον Οκτώβριο και η ψηφοφορία θα γίνει τον Νοέμβριο. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι το σημείο 6. Η εδώ είναι ο συνάδελφος Σαλβατόρε Γιακολίνο. Εδώ μιλάμε για το μέσο χρηματοδοτική στήριξη σε αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματο και διαχείριση κρίσεων. Ας ακούσουμε και πάλι την παρουσίαση της Επιτροπής και κατόπιν να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το θέμα που συμπεριλαμβάνει δύο νομικά μέσα, το ε, μέσο για την αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση κρίσεων, που είναι αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, και κατόπιν έχουμε τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις το οποίο θα είναι το επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη, το υπαριθμόν 7 στη μερίσια διάταξή μας σήμερα. Έχουμε λοιπόν σήμερα συζήτηση για την αστυνομική συνεργασία, τα δύο προγράμματα που έχουμε για το διάστημα 2007-2013 για την καταπολέμηση του εγκλήματος ε, και θα ακούσουμε την Κομισιόν, την Προεδρία και κατόπιν τον εισηγητή μας, κύριο Γιακολίνο. Θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σίφερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Το μέσο για την αστυνομία στα πλαίσιο του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης είναι το μικρότερο από τα δύο αυτά μέσα. Είναι αρκετά μικρότερο από το μέσο για τα σύνορα. Ένα δισεκατομμύριο προβλέπεται για την επταετία στο μέσο αυτό και ε, μπαίνουμε σε νέους τόπους με το μέσο αυτό, σε αντίθεση με τα ταμεία αλληλεγγύης, ε, τα οποία μπορούν να βασιστούν σε υπάρχοντα μέσα που υπάρχουν ε, από το 2005 και μετά. Αυτό δεν ισχύει για τον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και της καταπολέμησης του εγκλήματος. Καταλαβαίνετε την καινοτομία στα νέα στοιχεία της πρόταση αυτής, αν κοιτάξετε την υπάρχουσα κατάσταση και τα, αυτά που, μαθα, μάθαμε ε, από τις ελλείψεις της παρούσα κατάστασης. Σύντομα, λοιπόν να σας θυμίσω το πλαίσιο. Σήμερα στον τομέα της αστυνομία έχουμε δύο μικρά προγράμματα, το λεγόμενο ISAX και το SIPS ε, που έχουν να κάνουν με την ε, αστυνομική συνεργασία και την προστασία κριτικών υποδομών. Ε, τα οποία είναι μικρά, τα διαχειρίζεται αποκλειστικά η Επιτροπή, δεν καλύπτουν ε, το, την εξωτερική διάσταση, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Και τα δύο υπάρχοντα προγράμματα δεν συνδέονται ρητά με πολιτικές προτεραιότητες που συμφωνούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η ενδιάμεση αναθεώρηση των δύο αυτών μικρών προγραμμάτων ε, έχει ε, τονίσει αυτά. Υπάρχει λοιπόν αρκετά μεικτή, ε, υπάρχουν μεικτές απόψεις σχετικά με τα προγράμματα αυτά. Το 50% των ε, διαθέσιμων πόρων έχουν καταναμηθεί σε δύο μόνο ε, κράτη-μέλη, στο ένα σκέλος και στο ISAC, ε, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο. Τα, 50, τα 5 κράτη-μέλη αντιπροσωπεύουν το 50% της συνολικής αξίας των προγραμμάτων αυτών και το μισό των κρατών μελών δεν έκαναν καν το κόπο να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση η οποία σίγουρα δεν μπορεί να συνεφιστεί. Το νέο ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα να ευθυγραμμιστεί η ε, χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό με ε, καθιερωμένε αρχέ και κανόνες στον τομέα ασύλου μετανάστευση και συνόρων. Και γι' αυτό και στον τομέα της αστυνομίας. Θα προχωρήσουμε τώρα στη μοιρασμένη διαχείριση, αλλά επειδή είναι νέο αυτό για τις αρχές των κρατών μελών, αποφασίσαμε μόνο το 50% των πόρων να διατεθούν με κοινή διαχείριση. Το υπόλοιπο 50% θα το κρατήσουμε για ε, ενωσιακές δράσεις και προγράμματα. Ιδιαίτερα, όπως ακούσατε πριν. Στόχος είναι να ε, καλύψουμε και την εξωτερική ε, διάσταση που παίζει ρόλο και στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, της ασφάλειας ε, και θέλουμε να μπορούμε να καλύψουμε και επίγουσες δράσεις. Και αυτό είναι νέο στοιχείο. Έχουμε αυξήσει και την τεχνική βοήθεια σε σχέση με αυτά που έχουμε και που μπορούμε να ξοδέψουμε στα υπάρχοντα προγράμματα. Έχει αυξηθεί λοιπόν η τεχνική βοήθεια στα 8.000 ευρώ και το 5% του κομματιού ε, μοιρασμένης διαχείρισης ε, από τα κράτη-μέλη. Σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε όχι μόνο να βελτιώσουμε την οικονομική πλευρά της χρηματοδότησης στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας. Ε, κοιτάξαμε και τις ουσιαστικές δράσεις. Ε, κοιτάξαμε τις δράσεις οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν ή να διευρυνθούν ε, στο μέλλον και γι' αυτό σημαντικό είναι να θυμόμαστε το πλαίσιο πολιτικής. Από το 2010 και μετά έχουμε την ε, στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Υπήρχε μια ε, μακρά ανακοίνωση της Κομισιόν από τον Δεκέμβριο του 2010 όπου ε, αναφέρονται οι στρατηγικές προτεραιότητες από τις οποίες έχουμε επιλέξει πέντε προτεραιότητες τις οποίες έχουμε θέσει στο κέντρο του αστυνομικού αυτού μέσου. Έτσι λοιπόν δράσεις ε, που χρηματοδοτούνται είτε από τα ταμεία που διαχειρίζεται κεντρικά η Κομισιόν ε, είτε από τους πόρους που διαχειρίζονται ε, τα κράτη-μέλη στα πλαίσια προγραμμάτων υπό την μοιρασμένη διαχείριση. Προγράμματα από... θα μπορούν λοιπόν να χρηματοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό μέχρι 90% προγράμματα που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις πέντε στρατηγικές προτεραιότητες όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα 1 της πρότασης. Επίσης έχουμε διευρύνει και βελτιώσαμε, πιστεύουμε, ε, τον ε, κατάλογο επιλέξιμων δράσεων ε, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Νέο λοιπόν είναι στο προτινόμενο κείμενο ότι στο μέλλον θα πρέπει να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και δράσεις όπως είναι η εξέταση, η δοκιμή νέων τεχνολογιών. Αυτό δεν υπήρχε πριν και έχει οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις στο πρόβλημα ότι Έχουμε καλά αποτελέσματα ερευνών από το ε, πρόγραμμα πλαίσιο 6 και 7, αλλά δεν μπορούσαμε να τις ε, εφαρμόσουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια προεμπορική ε, δοκιμή των, των εφαρμογών αυτών και γι' αυτό το προσθέσαμε αυτό ως νέα δράση στο άρθρο για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις και προγράμματα. Επίσης η αγορά εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη ε, αυτή καθ' αυτή, μόνο ως ε, επιμέρους ε, κομμάτι προγραμμάτων που έχουν την ενίσχυση της εργασίας ως βασικό στόχο. Η ίδια η προμήθεια εξοπλισμού όμως δεν ήταν επιλέξιμη, ενώ στο μέλλον, για παράδειγμα στον τομέα των PNR θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τεχνικού εξοπλισμού, μέσων πληροφορικής. Θα είναι λοιπόν επιλέξιμα αυτά υπό ένα νέο μέσο. Για να σας αναφέρω δύο από τα πιο ε, σημαντικά παραδείγματα ε, όπου έχουμε διευρύνει τον κατάλογο των επιλέξιμων δράσεων. Όταν ε, μετακινούμαστε προς την μυρισμένη διαχείριση, προς την κοινή διαχείριση, ε, πρέπει να δώσουμε και οδηγίες σχετικά με την κατανομή των χρημάτων μεταξύ των κρατών μελών. Πώς θα γίνει η κατανομή των πόρων που θα είναι αντικείμενο κοινή διαχείριση, μοιρασμένη διαχείριση του 50%. Είμαστε βλέπουμε εδώ την πρώτη γενιά τέτοιων μέσων δεν υπάρχει προηγούμενο στο παρόν ε, πολιτεύσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έπρεπε λοιπόν ε, να βρούμε κάτι νέο. Σκεφτήκαμε λοιπόν ε, την χρήση αξιολόγησης κινδύνων και απειλών. Είναι δύσκολο να λάβει κανείς αντικειμενικές πληροφορίες και θα έπρεπε να βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά σε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι καλό σε περίπτωση οικονομικών μέσων τη στιγμή που το αντικείμενο είναι η κατανομή ε, πόρων μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό στραφήκαμε περισσότερο σε μετρήσιμους στόχους όπως ε, για παράδειγμα το τι θα πρέπει να προστατεύει τα αγαθά που θα πρέπει να προστατεύουν η αστυνομία ε, στα κράτη-μέλη, τον ε, πληθυσμό, τα εδάφη, τα εμπορεύματα ε, και τα λιμάνια και αεροδρόμια. Έτσι συγκεντρώσαμε αυτά τα πέντε κριτήρια τα οποία σταθμίσαμε και ανάλογα και προσθέσαμε και ένα πέμπτο κριτήριο, το οποίο είναι το ΑΕΠ, ώστε να φροντίσουμε η χρηματοδότηση να ωφελεί τα πιο φτωχά κράτη-μέλη, ώστε να αποφύγουμε οι ακριβές επενδύσεις στην ασφάλεια να γίνουν μόνο από τα κράτη-μέλη που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Φοβηθήκαμε ότι τα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να κάνουν τι επενδύσει αυτέ ε, θα ε, ε, αδικηθούν με μια κλίδα κατανομής που δεν θα λάμβανε υπόψη αυτό το κριτήριο. Αυτά λοιπόν είναι τα κριτήρια που επιλέξαμε και νομίζω ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στα έγγραφα που σας έχουμε μοιράσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα το Συμβούλιο, η Ιδανική Προεδρία. Κύριε Μέλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, προείπα, τον Ιανουάριο είχαμε μια συνάντηση με την Κομισιόν, όπου είχαμε μια παρουσίαση και σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Η προτινόμενη οδηγία αποτελεί καινοτομία και ετέθησαν πολλές ερωτήσεις προς την Κομισιόν σε εκείνη τη συνάντηση διευκρινιστικές ε, θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο και στα τέσσερα μέσα αλλά αυτό που αναφέρθηκε είναι στην νομική συνεργασία είναι όντως πραγματικότητα είναι το μικρότερο και σε επίπεδο χρημάτων φέσαμε να ξεκινήσουμε την πρώτη ανάγνωση αυτής της προτάσεως ε, όταν θα έχουμε κάνει περαιτέρω πρόοδο στην ε, υπόλοιπα ζητήματα. Ξεκινήσουμε την πρώτη ανάγνωση αρχές, ε, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Ε, επειδή λοιπόν η ομάδα του Συμβουλίου δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες της, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες προφορίες, αλλά επιβεβαιώνω πως Βλέπουμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο επί του θέματος και φυσικά είμαστε στην διάθεση του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε και τον εισηγητή τώρα, κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε την παρουσίαση της ε, Κομισιόν προηγούμενα και του Συμβουλίου τώρα για αυτό το σημαντικό ζήτημα, ότι το ταμείο αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτά που μας απασχόλησαν προηγουμένως. Πρόκειται για ένα μέσο για την ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, και της εθνικής συνεργασίας ε, που θα πρέπει να συνδέσει, συνδυάσει αυτές τις δραστηριότητε με τα αποτελέσματα που θα προέρθουν από την Επιτροπή κατά για την καταπολέμηση της μαφίας και την καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέθοδος ε, διαχείρισης η κοινή θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τα αποτελέσματα ως εκ τούτου η συνεχής ε, παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Τώρα για το αναλογία 5%, 5% ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη ε, και να μην οδηγηθούμε σε μια αποδυνάμωση του Ταμείου, κάτι για το οποίο θα επανέλθουμε φυσικά όταν ε, θα επιχειρηματολογούμε για αυτό το φάκελο. Το διεθνές έγκλημα επιβάλλει την συνεργασία είναι απαραίτητο να καθορίσουμε με βάση τον κατάλογο των στρατηγικών προτεραιοτήτων τις πέντε που συνοπτικά μας ανέφερε η Κομισιόν να γίνει λοιπόν μια ιδιαίτερη μνήα σε αυτές για τις οποίες ήδη μιλήσαμε και για τις οποίες θα πρέπει να αποδοθεί ένα, ένα πόρος συγκεκριμένος σαφής κάθε μία. Ένα... Κάτι ακόμα σημαντικό είναι, αφορά την διαχείριση της κρίσης των κρίσεων. Το συζητήσαμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ε, τα περιστάσεις στην ε, Λαμπεδούζα, διότι ε, δεν ε, μπορούσε κανείς να φύγει από το κέρας Αφρικής για να φτάσει και να ζητήσει άσυλο στην, ε, ούτε στη Σικελία ούτε στην Λαπεντούζα. Είχα προκύψει τότε το θέμα των ευθυνών. Ευθύνες ήταν... Ευθύνες μάλλον είχε και η Κομισιόν που θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερο θάρρος και αποφασιστικότητα το ζήτημα των έκτακτων καταστάσεων. Εκεί θα πρέπει να μπορούμε να παρεμβαίνουμε για να βρούμε μέσα τα οποία θα είναι ευέλικτα και άμεσης ε, εφαρμογής για να ενεργήσουμε σε συντονισμό με τα υπόλοιπα όργανα που έχουν αρμοδιότητες στο ζήτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Τώρα έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Κύριο Ταβάρη. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πρωτοδελικά Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα με αυτή τη λύση. Αν ήμασταν ομοσπονδιακό κράτος, λογικό είναι να έχουμε και αστυνομικές αρμοδιότητες. Από τη στιγμή όμως που δεν είμαστε ε, τέτοιο ομοσπονδιακό κράτος, ε, αισθάνομαι κάπως ε, περίεργα με αυτά τα αστυνομικά χαρακτηριστικά που κανονικά ανήκουν στα κράτη-μέλη. Αναφέρεται ο εξοπλισμός ή κάποιες δράσεις στα πλαίσια του PNR, του Μητρώου Επιβατών, θέματα που είναι επίμαχα ακόμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχω πρόβλημα το γεγονό ότι δεν είμαστε ομοσπονδιακό κράτο. Ούτε θα ήθελα όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε ένα υπερκυρίαρχο κράτο που θα αποκτά αστυνομικέ δραστηριότητε ή ερευνητικέ και διοκτικέ δραστηριότητε και θα εκπίπτει του κοινοβουλευτικού ελέγχου ταυτόχρονα. Γιατί αν θέλουμε ένα αντιστάθμισμα σε αυτή την αύξηση των αρμοδιοτήτων είναι η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν έχω πρόβλημα με, το... με την απόκτηση εξοπλισμού, αλλά δεν αναφέρονται πουθενά τα ατομικά δικαιώματα, η ιδιωτική σφαίρα, τα δικαιώματα του πολίτη και ούτω καθεξής. Ένα τμήμα των κονδυλίων αυτών, το 50% δηλαδή, που θα είναι το ποσοστό της Κρατική χρηματοδότηση. πολλές φορές τα κράτη-μέρη χρησιμοποιούν τα κοινοτικά κονδύλια για να κυκλώσουν τις πολιτικές τους ε, που δεν καταφέρουν να τι προβάλλουν σε ε, εθνικό επίπεδο. Ούτε ε, υπάρχει επαρκής έλεγχος των Εθνικών Κοινοβουλίων και δεν πιστεύω ότι θα μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχει καλά αυτέ τι ενέργειε. Γι' αυτό και αισθάνομαι κάπως άβολα με τι εξελίξει αυτέ. Σε ό,τι αφορά το 50% που θα διαχειρίζεται άμεσα απευθείας η Ένωση, για το, αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να ασκηθεί αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε για την απόκτηση εξοπλισμού, είτε για τα προγράμματα και τι προτεραιότητε τη Ένωση. Όλα θα πρέπει να ελέγχονται και να δίνεται το πράσινο φω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι και τι πολιτικέ ελευθερίε και τα δικαιώματα του πολίτη. Για να είμαι λοιπόν απόλυτα ειλικρινής, δεν είμαι και πολύ ενθουσιώδης ε, με την εισαγωγή του αντίθετου, αντίστροφου κανόνα του ΑΕΠ για το μέσο αυτό. Πιστεύω ότι αξίζει να χρηματοδοτήσουμε σε επίπεδο 90% κάποια προγράμματα των κρατών μελών, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον κάποιες ρήτρες σε ό,τι αφορά την, τις επιδόσεις των χωρών για την αξιοπιστία των ερευνών τους, για την ακαιρεότητα της αξιολόγησης των αστυνομικών δυνάμεων και φυσικά και μια αξιολόγηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Η εξασφάλιση των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Κρίμα που γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή, γιατί απουσιάζουν πολλοί από τους ενδιαφερομένους στην αποστολή στην Ουάσιγκτον, αλλά πιστεύω ότι θα, καλό θα ήταν να συνεχίσουμε τις συζητήσεις πάλι παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε άλλες συνεδριάσεις γιατί το γεγονό ότι αυτό το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης έχει πιο ε, περιορισμένο προϋπολογισμό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει λιγότερο ίσα ίσα γιατί τα ουσιαστικά του σημεία είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες. Δεν ζήτησε άλλος κανένα το λόγο. Οπότε επανερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και στο τέλος ο εισηγητής μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ε, διορθώσω μια παρανόηση. Το γεγονός ότι έχουμε συμπεριλάβει νέες δράσεις στον κατάλογο των επιλέξιμων δράσεων δεν σημαίνει ότι μπορούν απλά να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη χωρί να χρειαστεί να ασχοληθούν με τίποτα άλλο. Οι δράσει αυτέ θα πρέπει να πλαισιώνονται από εθνικά προγράμματα, από πολυετή προγράμματα, όλοι οι κανόνε που αφορούν τον προγραμματισμό και την εφαρμογή που αναφέρονται στον οριζόντιο κανονισμό ισχύουν και για το μέσο αυτό για την αστυνομία. Και δεύτερον, αν διαβάσετε το άρθρο 4 το οποίο περιέχει τον κατάλογο των ε, συνηθισμένων δράσεων, ε, θα δείτε ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους στο άρθρο 3 και τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από ό,τι βλέπω, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επενδύσουν τα χρήματα όπου θέλουν. Θα πρέπει να συνδέονται με τις πολιτικές προτεραιότητες, όπως για παράδειγμα ένα πιθανό μελλοντικό σύστημα ή ένα που να αποτελεί, ε, για τις πληροφορίες επιβατών δηλαδή, ε, ή να ε, συνδέονται με κάποια συμφωνημένη υποδομή. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Γιακολίνο, θέλετε να ολοκληρώσετε. Δεν έχω να πω πολλά περισσότερα, τα έχουμε πει ε, θα υπάρξει λοιπόν και μια, μια νέα συζήτηση. Περιμένω τις διάφορες ε, σύμβολες των συναδέλφων. Ε, αφήνω τον πρόεδρο τώρα να μας πει για το χρονοδιάγραμμα κλπ. Για μια ακόμα φορά θα σας υπενθυμίζω όπως και για τα προηγούμενα ζητήματα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρήσουμε εργαστήρι τον Απρίλιο Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε την έκθεση, προθεσμία καλά τροπολογιών τον Ιούλιο, εξέταση των τροπολογιών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και η ε, προσανατολική ψηφοφορία τον Νοέμβριο. Σημείο 8 της ίδιας ε, φύσης Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια, Εξωτερικά Σύνορα και θεωρήσεις εισηγητής ο συνάδελφος Μαριάν Ζαν Μαρινέσκου. Βρίσκεται στην αίθουσα. Όχι, είναι έξω από την αίθουσα. Παρατηρείτε. Μόλις επανέλθει θα ξεκινήσουμε. Κύριε Μαρινέσκου, ναι, ήρθατε. Ε, εσείς φταίτε, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ρώτησαν να πληροφορθούν σχετικά με τι συμβαίνει με την έκθεσή σας. Τώρα, αυτό το μέσο φορά μια ε, επέκταση του Σέγγεν Έχουμε την κυρία Μπελίντα Πάικ από την Κομισιόν. Μετά θα ακούσουμε την Δανική Προεδρία και εν τέλει τον εισηγητή μας, κύριο Μαρνέσκο, κυρία Πάικ. Ευχαριστώ. Το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα ενιαίο ταμείο, αλλά για νομικούς λόγους καλύπτει δύο μέσα. Πάντω, στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης, τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν εθνικά προγράμματα για να καλύψουν και τις δύο πτυχέ του Ταμείου εσωτερική ασφάλεια. Και τα εξωτερικά σύνορα διαχείριση των σύνορων είναι πολύ σημαντικό θέμα της Στρατηγική Ένωσης. Στόχος του Ταμείου αυτού είναι η διαχείριση των σύνορων ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασία των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα ομαλή διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα με βάση το κοινοτικό κεκτημένο για τα σύνορα. Και δεύτερος στόχο είναι η στήριξη της κοινή πολιτικής θεωρήσεων και εξασφάλιση της μεταχείρισης υπηκών χωρών και ε, διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Έχουμε μεγάλο προϋπολογισμό, 3,2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια από αυτά εμπίπτουν στην κοινή διαχείριση. Ένα τμήμα είναι πάγιο ποσό με βάση κριτήρια που σχετίζονται με τους στόχους, δηλαδή ε, με, με αντικειμενικούς συγγνώμη, παράγοντες όπως είναι η έκταση των συνόρων και ε, λεπτομεριακές πληροφορίες που θα υποβληθεί. 1,2 δισεκατομμύρια ε, κατανέμονται πάγια, με βάση μια πάγια βάση. Θα πρέπει κάθε κράτος να έχει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χώρα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική της τοποθεσία, γιατί θα έχει κάποια λειτουργικά κόστη που απορρέουν από την εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν. Ήδη στην έναρξη της του, της περίοδου προγραμματισμού δόθηκαν 450 εκατομμύρια στα κράτη-μέλη που συνιστούν μια ελαστική βάση. Εξαρτάται βέβαια σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη θέλουν να εφαρμόσουν τα μέτρα που προσδιορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού είτε για τη συνεργασία των προξενείων, είτε για κάποιες κοινέ επιχειρήσεις της Frontex. Θα επανέλθω σε αυτό εντός ολίγου. Επίσης, προβλέπεται 350 εκατομμύρια και μια ενδιάμεση αναθεώρηση. Με βάση την κοινή ε, διαχείριση προβλέψαμε 150 εκατομμύρια ευρώ για τα ιδιαίκα καθεστώτα ε, διαέλευσης με βάση τις ιδιαιτερότητες της Λιθουανίας. 2,2 δηλαδή σε εκατομμύρια με την, στην κοινή διαχείριση. Η διαχείριση των το, ταμείου γίνεται με κεντρικό τρόπο αλλά έχουμε και μία προσημείωση για το πακέτο α, έξυπνα σύνορα με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποβληθεί πριν το καλοκαίρι για ένα σύστημα εισόδου-εξόδου και ένα πρόγραμμα καταχωρημένων επιβατών. Θα θυμάστε ότι είχαμε υποβάλει μια ανακοίνωση με το περιεχόμενο αυτό το, φθινοπο, το φθινόπωρο και έγινε και μια διάσκεψη στα πλαίσια της ε, Δανικής Προεδρίας στην Ολλανδία παρουσία πολλών ευρωβουλευτών και της κυρίας Κέλλερ και οι νομικές προτάσεις θα υποβληθούν πριν το καλοκαίρι. Πάντως ήδη έχουμε προσημειώσει από το Ταμείο για την Ιστορική Ασφάλεια το Τμήμα για τα Εξωτερικά Σύνορα 1,1 δις για τις δράσεις στα κράτη-μέλη σε κεντρικό επίπεδο και για τη διαχείριση του συστήματος σε κεντρικό επίπεδο. Και μας μένουν 270 εκατομμύρια για κοινοτικέ δράσεις και άλλες λοιπές δράσεις. Θα σας επισημάνω κάποια στοιχεία του Ταμείου, του Ταμείου για την Εσωτερική Ασφάλεια, Εξωτερικά Σύνορα και Θεωρήσεις. Είναι ευρύτερο αυτό το Ταμείο από το ισχύον Ταμείο για, την, για τα Σύνορα και καλύπτει όλες τις πτυχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των σύνορων με βάση το τετραπλό μοντέλο πρόσβασης που περιλαμβάνει ε, συνεργασία με τρίτες χώρες, έλεγχο των συνόρων και κάποια μέτρα στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης. Μία σημαντική καινοτομία του ταμείου αυτού είναι ότι μέχρι 50% δηλαδή το πολύ τα μισά κονδύλια που εμπίπτουν στην κοινή διαχείριση των κρατών μελών μπορούν να δοθούν για επιχειρηματική λειτουργική στήριξη για την πρόθεση της διαχείρισης των συνόρων, για την ανάπτυξη μια κοινή πολιτικής θεωρήσεων και για την εφαρμογή συστημάτων ε, τεχνολογίας και επικοινωνιών όπως το ΣΥΣ, το ΒΙΣ και τα προγράμματα στο μέλλον καταχωρημένων επιβατών. Βέβαια αυτό εξαρτάται από τη συμμόρφωση των ενδιαφερομένων κρατών μελών με το κεκτημένο του Σέγγεν και ιδιαίτερα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 που προβλέπει ότι η λειτουργική επιχειρηματική στήριξη προσφέρεται μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των κρατών μελών με το κεκτημένο για τα εξωτερικά σύνορα και τι θεωρήσει και η συμμόρφωση με τι προδιαγραφέ και τι κατευθυντήριε γραμμέ για τα σύνορα και τι θεωρήσει. Η αιρεσιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και για τον εισηγητή και αναμένω συζήτηση για το θέμα αυτό ένα τρίτο χαρακτηριστικό του Ταμείου για την εσωτερική ασφάλεια, εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις σχετίζεται με τη διαχείριση, διακυβέρνηση του Σέγγεν. Το είπα αυτό και προηγουμένως απαντώντας τον κύριο Μέλντερ. Το Ταμείο θα στηρίξει κάποιους μηχανισμούς ε, στήριξης και παρακολούθησης και αξιολόγησης, χρηματοδοτώντας κάποιες ε, επιχειρήσεις ε, και τεχνική αρρωγή, εξετάζει αιρεσιμότητα σε ό,τι αφορά τη που είναι σημαντική, δηλαδή συμμόρφωση με το κεκτημένο του Σέγγεν και επιτρέψει στα κράτη-μέλη επαναπροσδιορισμό των πόρων, των κονδυλίων, εφόσον τα πορίσματά τους από την αξιολόγηση του Σέγγεν δείχνει κάποιες αδυναμίες στη διαχείριση των σύνορων. Άλλο σημείο σημαντικό αφορά την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Eurosort και με βάση το ταμείο αυτό θα χρηματοδοτήσουμε εισαγωγή και λειτουργία του Eurosol, του συστήματος δηλαδή επιτήρησης των συνόρων και θα παράγουμε, παράσουμε συνδρομή στα κράτη-μέλη. Πέμπτο στοιχείο της πρότασης είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό δυναμικό του οργανισμού Frontex. Ε, με βάση τον αναθεωρημένο κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου του 2011. Τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν συμπληρωματικά κονδύλια με βάση την κοινή διαχείριση, αναφέρθηκα σε ελαστικό τον ποσό, σε ό,τι αφορά την αγορά κάποιων μέσων που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων με τον Frontex καταρτήσουμε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το τι εξοπλισμός απαιτείται για τις κοινέ αυτές επιχειρήσεις με το Frontex. Τέλος, το γεγονός ότι είναι ελαστικά τα ποσά δεν παρέχει ενάβσματα στα κράτη-μέλη και προβλέπει και δυνατότητα χρηματοδότησης για προξενική συνεργασία τουλάχιστον μεταξύ δύο χωρών μελών προκειμένου να γίνεται ε, διαχείριση των θεωρήσεων σε ένα κοινό κέντρο υποβολή αιτήσεων, για παράδειγμα. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την συνεργασία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ε, των εξωτερικών συνόρων. Αυτά και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις. κυρία Μίλε τώρα από το Συμβούλιο, την Δανική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και στο ζήτημα αυτό μπορεί να είμαστε ιδιαίτερα σύντομοι. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και με την Κομισιόν. Τον Ιανουάριο έγιναν όλα αυτά. Όσο για την άλλη πρόταση, όσο γυρνούν κράτη-μέλη ε, με ευμένω υποδέχονται την πρόταση. Η πρώτη ανάγνωση τη προτάσεω θα ξεκινήσει αύριο. Και αυτό είναι ένα λόγο για τον οποίο δεν μπορώ να σα πω τίποτα παραπάνω αλλά για την τελευταία φορά, για σήμερα τουλάχιστον, σας επιβεβαιώνω την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και τον εισηγητή. Ας ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαρινέσκου, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η εφαρμογή του κανονισμού στηρίζεται στον διάλογο που η Κομισιόν θα έχει με τα κράτη-μέλη με κάθε ένα από αυτά και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποια είναι η προθεσμία για τον διάλογο αυτό. Διότι δεν αναφέρει στον κανονισμό κάποια προθεσμία. Υπάρχει μια προθεσμία για τα κράτη-μέλη εντός τριών μηνών από το πέρας του διαλόγου θα πρέπει να υποβάλουν ένα εθνικό πρόγραμμα. Αλλά πουθενά δεν είδα να αναφέρεται κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάποια καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του διαλόγου. Επίσης να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, αντιλαμβάνεται αυτά που αναφέρονται στο εθνικά προγράμματα για τα ΕΦΗ σύνορα, e Eurosur και την κανονισμό για την αξιολόγηση του Schengen. Όλα αυτά βρίσκονται στα ασκαριά και πιστεύω ότι η ανάπτυξη του ΣΥΣ 2 επηρεάζει τα εθνικά προγράμματα. Πώς λοιπόν η Κομισιόν τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα και με τη χρήση των πόρων. Και τέλος, πώς γίνεται η κατανομή των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία εθνικών προγραμμάτων, με τι κριτήρια γίνεται η κατανομή των πόρων. Υπάρχει μια ενδιάμεση αναθεώρηση όπου κάποιες διορθώσεις θα μπορέσουν να γίνουν, αλλά τα βασικά κονδύλια έχουν αποδοθεί ευθύ εξ αρχή. Δεν θέλω να γνωρίζω ποια ήταν τα κριτήρια με βάση τα οποία δόθηκαν τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Κύριος Ένσιο έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω την πρωτοβουλία αυτή για το μέσον για τις θεωρήσεις μετά το 2014. Όπως είπε η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ε, μια βασική λειτουργία σε επίπεδο ενωσιακό γιατί αυτό αφορά και τα σύνορα Σέγγεν, όχι μόνο τα εθνικά σύνορα. Χρειάζεται λοιπόν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Να τονίζω όμως ότι αυτή η στήριξη θα πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Εξ αυτών η σημαντικότερη είναι η τήρηση του κεκτημένου Σέγγεν. Γι' αυτό και συμφωνώ με τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η Κομισιόν θα χρειαστούμε αυτόν τον μηχανισμό αξιολόγηση και την σωστή διαχείριση της ε, ζώνης ε, Σέγγεν, διότι πρέπει να αποκατασταθεί η πλήρη εμπιστοσύνη ανάμεσα στο ε, μέλη που συμμετέχουν στο σύστημα Σέγγεν. Ο κύριος Μαρινέσκου, ο εισηγητής μας, και αυτός ε, είχε τις ε, ίδιες ε, με μένα ιδέες και επιθυμώ να υπογραμμίσω ένα σημαντικότατο ζήτημα το οποίο θα γίνει δεκτό από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν. Νομίζω ότι το 1,1 δις ευρώ που προβλέπονται για τα ευθύ σύνορα είναι μια σωστή απόφαση, αλλά οι προτεραιότητες μας τώρα δεν είναι μόνο το σύστημα εισόδου-εξόδου ή το σύστημα ARD. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει ακόμα να διαπραγματευόμαστε για το θέμα των ευφύων συνόρων μέχρι ότου δεν οριστικοποιηθούν οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Μιλάω για το ΣΥΣ2, το πακέτο Σέγγεν, το πακέτο ασύλου, ε, αλλά και το ζήτημα της, ε, του πακέτου που αφορούν την νόμιμη μετανάστευση. Μαζί με την κυρία, κυρία Κέλλερ συμμετείχαμε σε διάσκεψη για τα ευφύ σύνορα στην Κοπενχάγη. Τέλος, δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Πρώτον, ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία κατανείματε τα κονδύλια για κάθε κράτος μέλος, διότι στην πρόταση αναφέρεται ότι περίοδο 2010-2012 Ε, αυτή μάλλον η περίοδος θα είναι η περίοδος αναφοράς. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάποια στοιχεία όπως η επέκταση των εξωτερικών συνόρων ή και τον αριθμό των ε, προσώπων που ε, διασχίζουν τα σύνορα αυτά και το ζήτημα των εσωτερικών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Και όταν ε, προσωρινά ε, αποκαθίστανται αυτά τα σύνορα για λόγους ε, ελέγχου της κυκλοφορίας, πιστεύετε ότι θα πρέπει το Ταμείο αυτό να προστατεύει την διακίνηση διαμέσου των σύνορων στην περιοχή Σέγγεν, κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές από τις ερωτήσεις που έθεσα για τις γενικές διατάξεις ισχύουν και εδώ. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία, ποιος συμμετέχει σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο κλπ. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Ένσιου, εάν θέλουμε να δώσουμε ένα σωρό χρήματα ε, σε κάτι για το οποίο δεν έχουμε καν ξεκινήσει να νομοθετούμε, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό όσον αφορά την πολιτική συζήτηση. Αλλά για να δημιουργηθεί άλλη μία μεγάλη βάση δεδομένων τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν θα τεθεί ποτέ σε λειτουργία, αυτό είναι δύσκολο πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει για το πρόγραμμα EURES, ε, διότι θα είναι τόσο ακριβώς ο εξοπλισμός που θα ξεπερνάει οτιδήποτε συμπεριλάβουμε τώρα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό είναι άλλο ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα, μιλάτε για κάποια πιλωτικά προγράμματα για να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες που θα χρηματοδοτηθούν ε, μέσω του ε, ISF και μπορείτε να μου πείτε τι προγράμματα είναι αυτά και επίσης θα ήθελα να ξέρω αν χρήματα από το ISF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το κόστος των κρατών μελών για τα σύνορα. Μπορούν δηλαδή να πάρουν χρήματα από το ISF γι' αυτό ή θα γίνουν ε, όλα όσα αφορούν τα ΕΦΗ e σύνορα ε, με άμεση διαχείριση των χρημάτων. Ο συνάδελφός σα είναι ε, ακόμα και γι' αυτό θέλω να δράξω την ευκαιρία να ρωτήσω σχετικά με τη Γενική Διάταξη στο άρθρο 42 που λέει ότι παραβίαση ε, κοινοτικού, εθνικού ή ε, θα οδηγήσει σε κυρώσεις ε, με κάποιες προϋποθέσεις και αναφέρονται προϋποθέσεις η επιλογή προγραμμάτων υπό το εθνικό πρόγραμμα ή αν η παραβίαση έχει επηρεάσει τον, το, το ποσό ε, που θα πρέπει να επιστραφεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Μία σύντομη παρατήρηση. Ε, διότι σίγουρα θα κοιτάξουμε το θέμα αυτό και στην ε, ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού που είναι συναρμόδια. Υπάρχει ένα σύστημα εισόδου-εξόδου, ένα μεγάλο πρόγραμμα. Θα χαιρόμουν πολύ αν ξεκινούσε να λειτουργεί το ΣΥΣ 2 πρωτού να προχωρήσουμε στο επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει καταρχήν να διαπιστώσουμε, να αποδείξουμε ότι αυτό που έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χωρίς άλλες καθυστερήσεις, δυσκολίες ε, και ε, άλλα προβλήματα. Και επίσης ε, σημαντικό είναι να μπορούμε να αντιδρούμε άμεσα σε προβλήματα, σε ανάγκες. Ε, η Frontex δεν είναι πάντα διαθέσιμη όταν ε, είναι απαραίτητη. Νομίζω ότι έχει πολύ σημαντικό ε, ρόλο η Frontex και θα πρέπει να μπορεί να αντιδράει όταν της ζητείται αυτό και όχι μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε προβλέψει πριν από ένα ή δύο χρόνια. Άλλωστε αυτή είναι η δυο χρονια αλλωστε τι ειναι η δυναμη της Frontex να μπορεί να βοηθάει γρήγορα σε περιπτώσεις απρόβλεπτες και μη προγραμματισμένε. Θα πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα αυτή για τη Frontex και να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, η κυρία Πάικ. Thanks um, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο που έχει να κάνει με τη σημασία της Frontex. Ε, χθες και σήμερα ε, είχε συνάντηση ε, το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Frontex στη Βαρσοβία για να συζητήσει πώς μπορεί να αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την υιοθέτηση του προϋπολογισμού του 2012 προέβλεπε και τροποποίηση για την Frontex ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα της καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό. Η Κομισιόν δεν έχει λάβει ακόμα επίσημα αυτή την τροπολογία του κανονισμού. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω όμως ότι ο στόχος είναι να ε, τροποποιηθεί η δομή του κανονισμού ώστε οι ε, αξιωματικοί που ε, είναι επικεφαλής ε, των διαφόρων επιχειρήσεων όπως αυτός για τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι πράκτορες της υπηρεσίας και όχι, των κρατών, και όχι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Σίγουρα πάντως συζητήθηκε πολύ το θέμα αυτό χθες. Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω σε κάποια από τα άλλα θέματα η προθεσμία για τον πολιτικό διάλογο. Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσουμε εδώ, διότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τον πολιτικό διάλογο προτού να υιοθετηθούν οι ε, κανονισμοί. Ε, σας είπα ότι είναι πρόθεση της Κομισιόν να εκδώσει ανακοίνωση που να περιγράφει τη διαδικασία και τις προσδοκίες από τον πολιτικό διάλογο. Δεν μπορώ όμως να σας πω συγκεκριμένα πότε θα γίνει αυτό, διότι όλα εξαρτώνται από το πότε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα εγκρίνουν τους κανονισμούς. Ε, σαφές είναι ότι είναι προς συμφέρον όλων τα κράτη-μέλη να έχουν εθνικά ε, προγράμματα για το διάστημα 2014-2020, ε, το 2014 κατά προτίμηση ε, του χρόνου λοιπόν το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο μάλλον θα έχουμε εντατικό πολιτικό διάλογο με τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το, την κατανομή των πόρων. Στο παράδειγμα 1 του κανονισμού αναφέρονται τα ποσά που είναι η βάση των εθνικών προγραμμάτων για τα κράτη-μέλη. Και έχουμε πάρει τα ποσά για το διάστημα 2010-2012 ε, στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Και να σας θυμίσω ότι τα τέσσερα κριτήρια για την κατανομή των χρημάτων στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων είναι ε, υπάρχει στάθμιση, ε, είναι 30% για, τους, για τα εξωτερικά χερσαία σύνορα, 35% για τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, 20% για ε, αεροδρόμια και, και 15% ε, για το, τα προξενικά γραφεία. Οι λεπτομέρειες υπάρχουν στο Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα. Αυτή είναι η βάση λοιπόν για ε, την κατανομή των πόρων αυτών. Όσον αφορά το θέμα των ευφυών συνόρων, η Κομισιόν θεώρησε ότι είναι απαραίτητο δεδομένου του ότι στο περσινό πρόγραμμα εργασίας μας και στο φετινό λέμε ότι η Κομισιόν θέλει να προωθήσει το θέμα των εφιών συνόρων σε ανταπόκριση ε, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πέρσι που μας καλούν να ε, κινηθούμε γρήγορα και να παρουσιάσουμε ε, πρόταση. Ήδη πέρσι σε ανακοίνωσή μας το φθινόπωρο περιγράψαμε ε, το πεδίο εφαρμογής ε, των ε, προγραμμάτων εισόδου-εξόδου και για τους ταξιδιώτες. Και περιγράψαμε σε μία διάσκεψη την χρηματοδότηση και την ανάπτυξη αυτών και σε εθνικό και σε κεντρικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση θα γίνει από αυτό το 1,1 δισεκατομμύριο και κατόπιν και επίσης ε, στο, άρθρο 15 ε, περιγράφεται ο μηχανισμό. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν μέρο των εθνικών τους ε, προγραμμάτων από το Ταμείο αυτό για να χρηματοδοτήσουν το εθνικό κομμάτι. Αυτό όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα. Σημειώνω τι παρατηρήσει ε, που ακούστηκαν θα βρει να περιμένουμε να δούμε πώ λειτουργούν τα άλλα συστήματα προτού να προβλέψουμε νέα. Δεν θα πρέπει να αποτιμάμε τα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί. Το σύστημα πληροφόρηση ε, θεωρήσεων ε, λειτουργεί καλά. Το, Schengen, το σύστημα πληροφόρησης Schengen ε, μας έχει διδάξει πολλά σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων και νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα είναι ότι δεν ξεκινάμε την ανάπτυξη μέχρι να συμφωνήσουμε τι θα κάνει το σύστημα και γι' αυτό ο προγραμματισμός μας θα προβλέπει Εφόσον ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίσουν για την ύπαρξη των συστημάτων αυτών, η ανάπτυξη θα ξεκινήσει μετά την υιοθέτηση των σχετικών κανονισμών. Εάν λοιπόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, συμφωνήσουν το 2014, θα έχουμε την ανάπτυξη κατά το 2015 ε, έως 2017 και κατόπιν θα ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος από το 2018. Και επειδή και επειδή είναι πολύ σημαντική αυτή ε, η δέσμευση αναγνωρίζουμε ότι οι συζητήσεις και για τις προτάσεις και για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ε, συνδέονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά. Ο κύριος Μαρινέσκο επίσης ρώτησε σχετικά με το πώς λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις εξελίξεις ε, στο ε, σύστημα πληροφόρησης Schengen, εισόδου και εξόδου κλπ. Η χρηματοδότηση που παρέχεται στα κράτη-μέλη από τα εθνικά προγράμματα γίνονται με βάση τις προβληπόμενες εξελίξεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες πάνω στις διάφορες πτυχές του συστήματος Eurosol. και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δούνε τι είδου χρηματοδότηση θα είναι απαραίτητη. Πιστεύουμε ότι η πρόταση που έχουμε κάνει είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να λάβει υπόψη το γεγονό ότι ελπίζουμε ότι θα γίνουν εξελίξει στο σύστημα διαχείριση Σέγγεν, στον κώδικα διαχείριση ε, στον κώδικα συνόρων Σέγγεν ε, και στην αξιολόγηση Σέγγεν. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο ε, έλεγχος των εσωτερικών συνόρων θα είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση. Ε, θα σημειώσατε ότι στο άρθρο 4.4 λέμε πολύ συγκεκριμένα ότι δεν ε, είναι επιλέξιμα τα σύνορα. Όπου επανεισάγονται έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, ε, αυτό γίνεται σε προσωρινή βάση και για να καλυφθεί μια συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ε, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί επιπλέον χρηματοδότηση για αυτό. Οι αποφάσεις ε, που θα λαμβάνονται για την επανεισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα προποθέτουν και τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μπορούν να ε, ενημερώνουν σχετικά με τον αντίκτυπο για να μπορούν να επηρεάσουν τι αποφάσει αυτέ. Κύριε Μαρινέσκου, θέλετε να κλείσετε. Τίποτα ιδιαίτερο. Ε, προς το παρόν ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία και εκ των προτέρων ευχαριστώ για το Συμβούλιο για την ελπίζω μελλοντική αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μετά την, το σεμινάριο, το σχέδιο έκθεσης, ε, η προθεσμή για τις τροπολογίες, συζήτηση και ψηφοφορία θα ακολουθήσει το πρόγραμμα που έχουμε ορίσει και για τις προηγούμενες εκθέσεις που αφορούν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα τα επιμέρους θέματα που συζητήσαμε θα ακολουθήσουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9, αλλά το τελευταίο απογευματινό θέμα είναι το σημείο 8, οι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2013. Προβλέπεται η πρώτη ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Εισηγητή για τον Προϋπολογισμό του 2013, τον κύριο Τζοβάνι Λαβία. Our Σας καλωσορίζουμε θερμά κύριε Λαβία για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013 Μάλιστα θα υποβληθεί στις 25 Απριλίου. Αυτή είναι, αυτός είναι ο προγραμματισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η το σχέδιο γνωμοδότησης με τις προτεραιότητες μας για τον τριμερή διάλογο του Ιουνίου. δεν μπορούν να γίνουν χωρίς προηγούμενη πρώτη ανταλλαγή απόψε με το Γενικό Εισηγητή για τον Προϋπολογισμό, τον κύριο Λαβία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως ε, είπατε, στην τελευταία ολομέλεια κάναμε το πρώτο βήμα της μακράς διαδικασίας που μας οδηγεί στα τέλη του έτους ε, στην έγκριση του προϋπολογισμού για το 2013. Εγκρίναμε στην Ολομέλεια τις κατηδές γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2013 όπου συμπεριλαμβάνονται κάποιες γενικές πτυχές, κάποιες ώρε για το Κοινοβούλιο. Τι τις λεπτομέρειες όμως, αυτά που αφορούν ε, επιμέρου κεφάλαια του προπολογισμού θα ε, εξεταστούν ε, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου όπου προτίθεμε να φροντίζουν να εμπλακούν όλες οι κοινοβουλευτικές τροπές του Κοινοβουλίου για να έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και να μπορέσω σε εκ τούτου να εξετάσω τα επιμέρους κεφάλαια του προπολογισμού. Φυσικά θα έχω μια πολύ στενή επαφή και συνεργασία με όλους τους εισηγητές ε, για τις του Κοινοβουλίου, όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και από κοινού θα οικοδομήσουμε την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Δεν διαφεύγει το γεγονό ότι το 2013 ο προπολογισμό θα είναι ο τελευταίο ε, το, στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όπως καταλαβαίνετε είναι μεγαλύτερη προσοχή που αποδίδεται σε ό,τι φορά στις πληρωμές δεδομένου ότι τα προγράμματα τρέχουν και είναι απαραίτητη πόρη για τις πληρωμές σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός είναι και ο προϋπολογισμός ε, αναφορικά με τις προβλέψεις που κάνουμε μετά από το 2011 ε, όπου είχαμε σημαντικές δυσκολίες διότι το Συμβούλιο είχε θέσει κάποιους περιορισμούς ε, στις πληρωμές πολύ στενούς, κάτι το οποίο οδήγησε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς παράλληλα με τίματα από τα κράτη-μέλη για πληρωμές να υπάρξει λοιπόν μια μεταφορά πληρωμών από το 2011 στο 2012. Τα κράτη-μέλη λοιπόν μόνο το τελευταίο μάτι του 2011 ε, υπέβαλαν αιτήσει για πληρωμές στη τάξη του 16 δις Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάνω από 11 δις ε, θα πρέπει να καταβληθούν το 12, διότι μόνο 5 δισεκατομμύρια μπόρεσαν να καταβληθούν πριν από το τέλη του 11. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του έτους ε, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε την πρόοδο των πληρωμών για να αποφύγουμε το κλείσιμο του προπολογισμού για την επόμενη χρονιά να ενταθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε πέρυσι. προσέξαμε ιδιαίτερα δύο βασικές πτυχές επί των οποίων θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία. Πρώτα απ' όλα, ανάπτυξη και ε, μεγέθυνση ε, με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο, συγγνώμη, να εξετάσουμε, το ζήτημα, υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που άπτεται της απασχόλησης και σχέση με τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον νότο της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά θελήσαμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσίε επιχειρήσεις, διότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές που την τελευταία δεκαετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατόρθωσε να απορροφήσει το 85% της νέας ε, απασχόλησης. Στις μικροφύσεις επιχειρήσεις λοιπόν θα θέλουμε να αφιερώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Όλα αυτά φυσικά με αναφορά στα επιμέρους κεφάλαια του προπολισμού θα συζητήσουμε στο πλαίσιο του ημέρου διαλόγου και ζητώ από την Επιτροπή σας ε, μια ουσιαστική συνεργασία ε, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας. Ε, εξάλλου θα ήθελα να υπογραμμίσω και άλλη μια πτυχή. Το ζήτημα των πιλωτικών ε, προγραμμάτων για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου που είναι στοιχεία που θέλουν να ενεργοποιήσουν δραστηριότητες επί ζητημάτων που δεν καλύπτονται από μια γραμμή του προπολογισμού σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές ε, ε, δραστηριότητες θα φτιάξουμε ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο που θα μας επιτρέψει να υποβάλουμε αυτές τις πρωτοβουλίες προκαταρκτικά στην Εκτελεστική Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί ε, το, το, ο εφικτός χαρακτήρας τους Ανάλογα λοιπόν με το ότι έγινε πέρυσι, θα ζητήσουμε προκατακτικά από τις ε, αρμόδιες επιτροπές και άρα και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τις προτάσεις τους σε ό,τι φορά τις προπαρασκευαστικές ε, δράσεις ε, και τα πιλωτικά προγράμματα ώστε να μπορέσουμε να αποστείλουμε αυτές τις προτάσεις μέσα με τέλη Ιουνίου στην Εκτελεστική Επιτροπή έτσι ώστε να έχουμε μια αξιολόγηση προκατακτική αναφορικά με το εφικτό αυτών των προγραμμάτων. Και επί του θέματος αυτού θα ψηφίσουμε μετά τις θερινές διακοπές. Ε, ζητώ από την Κομισιόν και από τον εξειδικευμένο εισηγητή σας να συνεργαστούμε για να κλείσουμε στα τέλη του έτους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ώστε να μπορέσουμε να θα πάμε στον ε, τελική συζήτηση με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ε, ε, συναλλαγής να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για το πολιτισμό 2013. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Λαβία για αυτή την προσέγγιση που έχετε στο Πολιτισμό 2013. Γνωρίζουμε πως ε, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει ήδη διορίσει εισηγητή. Κύριε Γιακολίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Λαβία για την ε, συγκεκριμένη άποψη που μας ανέφερε όπου αναφέρονται ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά και απαιτήσει του προπολογισμού. Το είπε και ο κύριος Λαβία ε, όταν ε, στο Στρασβούργο εγκρίναμε την έκθεση ε, λιτότητα αλλά ανάπτυξη με μεγέθυνση. Εμείς θα εξετάσουμε το ζήτημα που εμπίπτει τι αρμοδιότητέ μα, δηλαδή το Ταμείο για την Ιστορική Ασφάλεια, το Ταμείο για το Άσυλο και την Μετανάστευση και όλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται τη δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα θέμα που άπτεται των πληρωμών, το είπε και ο συγγητή, πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ε, υπηρεσίε που αφορούν στην Επιτροπή μα, ε, και θα πρέπει να αξιολογηθούν ε, το κόστος και τα αποτελέσματα αυτών των υπηρεσιών χρειάζεται το 2013 να στηριχθούν οι δραστηριότητες που θα αφορούν την, την λειτουργία τους για μετά το 2013, δηλαδή για το 2014 να υπάρξει λοιπόν μια συνέχεια, διότι το 2014 θα είναι ε, η ημερομηνία έναρξη, μάλλον παράταση λειτουργίας. Μίλησαμε για ευθύνη, για αλληλεγγύη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες ε, στο Κοινοβούλιο και για να εγγυηθούμε ε, μάλλον θα πρέπει εμείς να εγγυηθούμε ως αρμόδια επιτροπή την ασφάλεια των πολιτών ε, αναφερόμενοι φυσικά και στις προπαρασκευαστικές δράσεις ε, και στα πιλωτικά προγράμματα όπως είπε ο κ. Δελαβία θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος των προτεραιοτήτων που θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν μέσα στο πνεύμα συνεργασίας ε, στην Επιτροπή μας και να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα που είπε και ο εισηγητής για να οδηγηθούμε σε έναν προπολογισμό ο οποίος θα ανταποκρίνεται τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο για αυτή την παρουσίαση. Ο κύριος Μπούζου Τίλ θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αλλά προτιμώ να μιλήσω αγγλικά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα σας, δι... διέφυγε ο ηρωνικός τόνος μου νωρίτερα όταν ψηφίσαμε ε, την ε, ανάθεση των, των ε, εκθέσεων. Ήταν όλοι παρόντος και τώρα που συζητούμε ε, τον προπολογισμό για ένα από τους πιο σημαντικού τομεί Ευρωπαϊκής Ένωση έχουμε μείνει τρει και ο κούκος για την ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Εισηγητή για τον προπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Λαδία που ήρθε για την ανταλλαγή απόψεων που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντική. Και είναι σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψε, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό του 1% του συνόλου του κοινοτικού προπολογισμού για τον τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων είναι ανεπαρκέστατο. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι το βασικό σχόλιο που θα πρέπει να συγκρατήσει από τη συζήτηση ο κύριος Λαβία. Η πολιτική δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων είναι από τι πιο σημαντικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αρμοδιότητα τη δική μα Επιτροπή και έχουμε κολλήσει μόλις στο 1% του κοινοτικού προϋπολογισμού για την πολιτική αυτή. Ανεπαρκέστατο επαναλαμβάνω το ποσοστό αυτό, ευτελέστατος και πολύ συρρυκνωμένος ο προϋπολογισμός. Κύριε Λαβία, οι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται για την αδικαιοσύνη, ενδιαφέρονται για τις εσωτερικές υποθέσεις, ιδιαίτερα για την αστυνομική συνεργασία, την τρομοκρατία, τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου και χρειαζόμαστε τους πόρους και τα κονδύλια για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε τις κοινέ μας πολιτικές προ όφελο των συμπολιτών μα. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω επίση, κύριε Λαβία, ότι όλο και μεγαλύτερο αριθμό οργανισμών εμπίπτει πια στι αρμοδιότητε τη Επιτροπή μα και οι περισσότεροι από του οργανισμού αυτού είναι νεοπαγεί. Τώρα ξεκινούν τη λειτουργία τους, ε, αρχίζουν και προσλαμβάνουν προσωπικό, βρίσκονται σε φάση ε, οργάνωσης και ρονταρίσματος ε, για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν την αποστολή τους. Χαίρομαι που ο κύριος Λαβία κατάγεται από τη Σικελία, γιατί σε θέματα μεταναστευτικά είναι σε θέση να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα που έχει η μεταναστευτική πολιτική, που επίσης ε, χρήζει σημαντικούς πόρους, χρήζει σημαντικών πόρων. Και θέλουμε ε, η Frontex, ο οργανισμός Frontex να ενισχυθεί ε, ε, στην αποστολή του και να περιλάβει και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, θα πρέπει να τον εφοδιάσουμε με τους απαραίτητους πόρους και όχι μόνο το Frontex αλλά και τους άλλους οργανισμούς. Εν λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ε, επαναλαμβάνω ότι ε, δεν είναι καθόλου τυχαίο που επιλέξαμε τον κύριο Γιακολίνο ως εισηγητή της γνωμοδότησης της ε, Επιτροπής μας, γιατί και αυτός κατάγεται από τη Σικελία και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία του με τον κύριο Λαβία, τον συμπατριώτη του θα αποβεί προς όφελος της Επιτροπής μας. Ναι, το σημειώνουμε όντως. Σχολιά, ε, λαμβάνουμε υπόψη το σχόλιο σας για το ηλεκτρικό, για την έκριθμη κατάσταση που ε, επικρατούσε στην Επιτροπή, ιδιαίτερα σε ό,τι το σχετισμό δυνάμεων και τη σύγκρουση δυνάμεων ε, για διάφορες ψηφοφορίες. Εκεί πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλο ηλεκτρισμό και αθρώα προσέλευση και μετά από τον πολύ ηλεκτρισμό καταλήγουμε στο blackout και στους ελάχιστους που έχουν απομείνει για να συζητήσουμε σημαντικά θέματα όπως ο προπολογισμό για το 2013. Σημειώσαμε λοιπόν το καυστικό σας σχόλιο. Ε, ζήτησαν το λόγο η κυρία Κέλλερ και η κυρία Χολμάιερ. Κυρία Κέλλερ, προηγήστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Το θετικό είναι βέβαια ότι μπορεί κανείς να θέσει περισσότερες προτεραιότητες ε, και να εκφράσει περισσότερες επιθυμίες όταν είμαστε λιγότεροι. Ε, συμμερίζομαι τη θέση σας ότι είναι λίγα τα χρήματα για τον τομέα εσωτερικών. Παρότι υπάρχει πραγματική ανάγκη ε, για πόρους. Θα πρέπει να δούμε που χρειαζόμαστε λεφτά. Θα πρέπει όμως ε, να ε, φροντίσουμε να μην ε, ξοδεύουμε υπερβολικά πολλά χρήματα σε διάφορου τομείς δημιουργούνται οι οργανισμοί, ε, ανατίθενται περισσότερες, περισσότερα καθήκοντα σε κάποιους υπάρχοντες οργανισμούς. Ε, έχουμε τον ΙΑΖΟ που ε, έχει μεγάλο αριθμό καθηκόντων. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τον οργανισμό αυτόν, καθώς και τον Ευρωπαίο Επόπτη για την προστασία των δεδομένων. Δεν θα πρέπει να υποχρηματοδοτούνται οι οργανισμοί αυτοί. Κάτι γενικό, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να γίνονται, νέες, να γίνονται καλές αξιολογήσεις προτού να προχωρήσουμε σε νέες πολιτικές. Δεν έχει νόημα να ε, δημιουργούμε νέα προγράμματα τη στιγμή που δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις των παλιών. Άλλο σημαντικό τομέα που θα μα αποσχολήσει αρκετό καιρό είναι ε, το Ταμείο Προσφύγων. Ε, δεν ε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση πολύ. Υπάρχει το δημοσιονομικό θέμα, υπάρχει το θέμα του προϋπολογισμού, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε με την τάση των οργανισμών, της Frontex και άλλων ε, να έχουν έναν προϋπολογισμό, αλλά στη μέση της, του χρόνου να ζητάνε ε, συμπληρωματικό προϋπολογισμό, κάτι το οποίο δεν περνάει από την Επιτροπή μας. Εμείς ε, καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό για έναν οργανισμό, μετά από ε, μισό χρόνο όμως ε, παίρνει περισσότερα χρήματα ο οργανισμός αυτός. Καλύτερα να έχουμε αποθέματα τότε. Οι οργανισμοί να μας λένε τι χρειάζονται. δεν είναι διαφανής ε, διαδικασία όταν έχουμε συμπληρωματικό ε, προϋπολογισμό εκ των υστέρων μετά από μισό χρόνο ή μετά από κάποιους μήνες. Ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, παρότι δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια μιας τέτοιας έκθεση για το προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χολμάιερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφε Τζοβάνι Λαβία, Όπως ε, είπε ο συνάδελφος Ποζουτήλ και η κυρία Κέλλα, Κέλλερ, ε, σημαντικό είναι να χρηματοδοτούνται επαρκώ οι τομεί αυτοί, πόσο μάλλον που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη στα θέματα αστυνομική συνεργασίας και μετανάστευση. Ε, θέλουμε με την Frontex ε, να προστατεύσουμε, σε συνεργασία με τη Frontex να ε, προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα. προστίθενται και νέοι τομεί όπου η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τουλάχιστον εξίσου καλή θέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εξετάζει θέματα που έχουν να κάνουν με το κυβερνοέγκλημα. Στο μεταξύ, υπάρχουν αρκετές καλές δυνατότητες να ενεργήσει κανείς αφενός προληπτικά, ε, αφετέρου δε να ε, να ε, μπορέσει να αντιμετωπίσει το, οργαν... το διεθνές οργανωμένο έγκλημα στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τις ζημιές ε, του κυβερνοεγκλήματος που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ε, να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να προσέξουμε το 2013 να ε, δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επαρκή μέσα ώστε να ξεκινήσει ε, τις προσπάθειες στον τομέα αυτών. Η Κομισιόν στις 28 Μαρτίου υπέβαλε σχετική ανακοίνωση και κατά τη διάρκεια του έτους 2013 θα πρέπει να ενεργήσουμε σωστά ε, διότι είναι τόσο σημαντικό το κόστος πια που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το θέμα αυτό, ούτε μπορούμε να το αφήσουμε στο κάθε κράτος μέλος. Πρόκειται για διεθνή δίκτυα και θα πρέπει να εξετάσουμε ε, τρόπους πρόληψης, έγκαιρης πρόληψης. διότι δυνατότητε δίνει το διαδίκτυο όχι μόνο σε αυτούς που το χρησιμοποιούν με λογικό τρόπο, αλλά και στους εγκληματίες. Ήθελα να το πω αυτό, διότι το θεωρώ σημαντικό και ε, στο πλαίσιο αυτών που έχουμε συζητήσει τον τελευταίο καιρό ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και για το εγκλήμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριος Μπρόγκς, τελευταίος ομιλητής, πριν ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Λαβία. Ευχαριστώ. Εγώ δυστυχώς θα παραφωνήσω σε σχέση με τους προλαλήσαντες. Ο κύριος Λαβία αναφέρθηκε στους οικονομικούς στόχους. Δεν είναι ε, επίκριση προς τον ίδιο, μορφή προς τον ίδιο. Δεν είναι εκείνος που αποφασίζει την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μορφή προς ε, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε η μεγέθυνση και ανάπτυξη αφενός και η απασχόληση αφετέρου ως σημαντικότερες προτεραιότητες ε, του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αν όντω ισχύει αυτό, τότε γιατί επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο νόμισμα που είναι υψηλό τίμημα για τι χώρε του Νότου και του εξαναγκάζει σε ανεργία και στασιμότητα, ενώ αν είχαν τα δικά του νομίσματα θα μπορούσαν να, να έχουν περισσότερε εξαγωγέ και ανάπτυξη. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κοινά επιτόκια για 17 χώρες. Γιατί δεν αφήνει ελεύθερες εμπορικές οικονομίες. Γιατί η Κίνα, ε, μια αναδυόμενη οικονομία με υποβαθμισμένο, υποτιμημένο ασκεμένα νόμισμα και χαμηλό ε, μισθολογικό κόστος, ε, ανταγωνίζεται τα κοινοτικά προϊόντα και έτσι υποβαθμίζεται η δική μας ε, βιομηχανία, ενώ οι λαθρομετανάστες ε, διεκδικούν ε, θέσεις απασχόλησης θερώντας από τους συμπολίτε μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής που παρέμειναν ακόμα στην αίθουσα και έθεσαν και κάποιες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Νομίζω ότι το... τα ποσά, τα κονδύλια που έχουμε στον προπολογισμό 2012 για τον δικαιοσύνη και εσωτερικές ποδές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, αλλά είναι σαφές πως αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς περιπέτεια και θα πρέπει να παραμείνουμε εντός του του ορίου του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και είναι σίγουρα δεν έχουμε πολλά περιθώρια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο <coughs> τα χρήματα που έχουμε ε, σύμφωνα με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό γνωρίζω πολύ καλά αυτό που ο κύριος ε, Μπουζουτήλ ότι έχουμε πολλές υπηρεσίες αλλά χρειάζομαστε και πολλά χρήματα για αυτές. Χρειάζεται όμως να χρησιμοποιήσουμε, επαναλαμβάνω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας με βάση το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε χρόνο για το συνθήσουμε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. <clears throat> Κυρία Κέλλερ και άλλα μέλη είπαν πως θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε άλλες γραμμές του προπολογισμού όπως το Ταμείο για τους ε, πρόσφυγες, ε, την ε, πολιτική μετανάστευσης πέρυσι είχαμε πετύχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στο Ταμείο των Προσφύγων και την μεταναστευτική πολιτική αφετέρου. Και βρίσκομαι εδώ για να σας ακούσω. Ακούσω τις προτεραιότητες της Επιτροπής και τι θα πρέπει να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τον τρόπο τα χρήματα. Άκουσα επίσης την ερώτηση για τον κύβερνο χώρο και την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι εθνικό. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πάνω στο ζήτημα. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, προς τον κύριο Μπρόνς. Το πρόβλημα που έθιξε είναι μεγάλο. Αλλά δεν είναι ρόλος του Γενικού Εισηγητή να απαντήσει σε αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε μια μεγάλη συζήτηση, μια μακρά συζήτηση περί αυτού και εγώ είμαι υπέρ. Αλλά δεν είναι πάντα δυνατόν να μιλάει κανείς κατά της Ευρώπης χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαβία για τη δουλειά που κάνατε και γιατί πρόκειται να κάνετε στο μέλλον. Ο εισηγητής μας για Κολίνα θέλει να προσθέσει κάτι. 30 δευτερόλεπτα πρόεδρο. Μετά από τα ίσια εγώ, κύριο Μπουζουτήλ είναι σωστό να ζητήσουμε περαιτέρω πόρους. Το 1% χορηγείται στους δραστηριότητες μας, αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα πώς δαπανήθηκαν οι πόροι στο παρελθόν και να φροντίσουμε ώστε οι πόροι του 2013 να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Τέλειωσα πρόεδρε, ευχαριστώ αυτά προς το παρόν. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε στις 9 μια τελική ανακοίνωση. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 θα παρουσιαστεί, όπως είπα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Απριλίου. Ο εισηγητή θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση, το σχέδιο γνωμοδότηση για τι προτεραιότητε για τον ε, τριμερή διάλογο στι 8 ε, Μαου. Θα τα πούμε αύριο.